Colleagues, Μπορούμε να αρχίσουμε κυρίες και κύριοι. Έτσι και θα γίνει. Ας αρχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσει ω προ την ημερήσια διάταξη. Όχι, φαίνεται, ε, εγκρίνεται λοιπόν ω έχει. Πρακτικά τη τελευταία συνεδρίασης της 22 Σεπτεμβρίου Υπάρχουν σχόλια. Um, Περιμένω σχόλια μέχρι το τέλος της ε, συνεδρίας, ενδεχομένως αλλιώς ε, θεωρείται ως ε, εγκεκριμένη. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Όπως ξέρετε, η... μπορεί να ακουστεί η συνεδρίαση αυτή μέσω διαδικτύου, εκτός από τη συνεδρίαση των συντονιστών. of the agenda. Και τα πρακτικά είναι διαθέσιμα. Running too fast. Um, Σημείο 4. Πρόεδρος των τριμερών διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν ε, δύο θέματα. Η, η ρύθμιση των διμερών συμφωνιών επενδύσεων που ισχύουν που ίσχυαν πριν από τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. Ξέρετε ότι είμαι εξορισμού εισηγητής. Έγινε μια σε μια συνάντηση που ήταν ιδιαίτερα θετική και ξέρετε ότι οι θέσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής έγινε απόλυτα, έγιναν απόλυτα σαφείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει ένα προσχέδιο κειμένου που θα είναι η βάση συμβιβασμού. Και ήδη έχει γίνει αυτό από την Επιτροπή, γι' αυτό νομίζω ότι κατά την προσεχή συνεδρίαση θα ασχοληθούμε με τροπολογία συμβιβασμού. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δύσκολο θέμα, αλλά παρά τις διαφορές μας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αρκετά γρήγορα. Ως προς το ICI, ξέρετε ότι είναι, υπάρχει μια διαδικασία συνδιαλλαγής σε σχέση και με ένα παρεμφερές ζήτημα από την ΤΕΒΕ και την Επιτροπή Εξωτερικών Υπόθεσεων για το ονομαζόμενο PCI, δηλαδή την συμμετοχή των ιδιωτών. Φτάσαμε. PCI είναι και όχι PSI. However... Έγιναν λοιπόν διαπραγματεύσεις και φτάσαμε σε μία συμφωνία, όμως τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου αμφισβητούν αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα αργότερα κατά τη σημερινή ημέρα και δεν μπορώ να προδικάσω το τι θα συμβεί, γιατί είναι μια ασύνηθης διαδικασία. Ο εισηγητής μας δεν είναι εδώ. Α. So let's give a second to Helmut Scholz to sign the list and I will ask him whether he Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να προσθέσετε κάτι ως προς τη διαδικασία συνδιαλλαγής για το ICI. Κασπάρη. Ναι, στα αγγλικά. Μόλις φτάνει ο συνάδελφος να τον αφήσουμε λίγο να εγκατασταθεί, να ξαναβρει τη ανάσα του. Θέλω να ρωτήσω, έχουμε τίποτα νέα ε, από το Συμβούλιο για τον κανονισμό που ψηφίσαμε για το ε, Made In την πρώτη ανάγνωση πριν από κάνα χρόνο νομίζω και δεν αντέδρασε το Συμβούλιο. Δεν έχει αρχίσει ακόμα ο τριμερής διάλογος. Θα με ενδιέφερε να έχουμε τίποτα νέα για αυτό το θέμα. Ε, από όσο γνωρίζω δεν υπάρχουν από το Συμβούλιο σε σχέση με το θέμα αυτό. Με συγχωρείτε που άργησα, αλλά ήρθα από κάποια άλλη συνάντηση. Σήμερα το πρωί είχα μία συνάντηση και θα ήθελα να πω ότι έγινε ο τελευταίος γύρος τριμερούς διαλόγου με, την, με τους συναδέλφους Γκέρενς, Λοχ, Μπίλερ και άλλων και εσείς συμμετείχατε και εγώ και στα συμπεράσματα θα ήθελα να πω ότι φτάσαμε σε προσωρινή συμφωνία σε σχέση με ένα πακέτο για τα δύο μέσα που μας απασχολούν μέσα στα πλαίσια αυτού του τριμερούς διαλόγου ACI Plus και ε, ECI, τον κανονισμό ECI. φτάσαμε σε μια συμφωνία ως προς το ICI, το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες, γνωρίζοντας ότι τα δύο θέματα, το άρθρο 16 και τις εξουσιοδοτημένες πράξεις, κατεξουσιοδότηση πράξεις καλύπτονται από μία δήλωση η οποία διέπει τον τρέχοντα κανονισμό με τις ε, προοπτικές του μελλοντικού μέσου μετά από την διετή πορεία μας. Άρα αυτή η μελλοντική προσέγγιση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, καλύπτεται από μία σύντομη δήλωση όπου και οι δύο πλευρές εκφράζουν τη θέλησή τους να εξετάσουν περαιτέρω το ζήτημα. Σε σχέση με το άρθρο 10 φτάσαμε σε μία προσθήκη, δηλαδή μία δήλωση, μία σύντομη δήλωση σε σχέση με τον αρχικό κανονισμό όπως προβλεπόταν στις διαπραγματεύσεις του Κοινοβουλίου. Και η δική μας διατύπωση κρατήθηκε ως διατύπωση η οποία θα επικρατήσει μετά από πρώτη και δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι επί του παρόντος συμβαδίζουμε με τα αποτελέσματα της ομάδας διαπραγματεύσεων. Σε σχέση με το DCI υπάρχει μια ομάδα διαπραγματεύσεων. Δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε. Σήμερα το απόγευμα προβλέπεται μια συνάντηση της ομάδας της αντιπροσωπείας και θα δούμε πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτό το ζήτημα. Αυτά μπορώ να σας πω επί του παρόντος. Συμφωνώ με τα συμπεράσματα του Helmut Scholz σε σχέση με το ICI, δηλαδή το δικό μας θέμα, τη δική μας πλευρά. Πάντα υπήρχε σύμπνια, τουλάχιστον μέχρι τούδε, και είχαμε συναντήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα με τις πολιτικές ομάδες άρα δεν έχουμε πρόβλημα να δεχτούμε τη συμφωνία. Είναι ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός, αλλά στις διαπραγματεύσεις δεν είμαστε 100% σίγουροι για την έκβαση του ζητήματος. Κατά τη δική μου άποψη και τη άποψη του εισηγητή θα πρέπει να δεχτούμε την ε, Συμφωνία Συμβιβασμού. Τώρα θα αποφανθεί η ομάδα διαπραγματεύσεων, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκπλήξεις. σε σχέση με την πρωτοβουλία που είχε αναλυφθεί. Αλλά δεν θα αποφασίσουμε εμείς εδώ. Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα αποφανθεί σήμερα το απόγευμα. Σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Προσθετικό πρωτόκολλο στην Ευρωμεσογειακή Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ισραήλ. Πρόκειται για μια συμφωνία, για ένα πρωτόκολλο σε σχέση με την αξιολόγηση συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανιών προϊόντων με το ακρονίμιο ΆΚΑ, Συμφωνία ΆΚΑ, σε σχέση με τα βιομηχανικά προϊόντα και την αποδοχή τους. Όπως ξέρετε, ανέλαβα πρόεδρος αργότερα, εισηγητής ενώ λέει ο πρόεδρος, διορθώνει, δεν την είχα αναλάβει, αναλάβει εξ αρχής αυτή την έκθεση, γι' αυτό περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις έτσι ώστε να σας υποβάλω ένα προσχέδιο έκθεσης. Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και στο τέλος της ανταλλαγής αυτής είτε θα έχουμε μία σαφή κατευθυντήρια γραμμή ή θα ψηφίσουμε για να γνωρίζω τις δικές σας θέσεις. και αυτή τη στιγμή δεν έχω χρονοδιάγραμμα, θα το έχω στο τέλος της συζήτησης. Λοιπόν, αρχίζει η συζήτηση, δεν έχουμε συζήτηση. Η κυρία Αντρικένε ζήτησε το λόγο. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και απλώς θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Συμβούλιο ενέκρινε αυτή τη συμφωνία το Μάιο του 2010 η συμφωνία αυτή αφορά την σύγκληση της ε, νομοθεσίας, των είπαμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την ανταλλαγή ιατρικών προϊόντων, όχι όπλων βεβαίως. Γι' αυτό θα ήθελα οι συνάδελφοι να επιταχύνουν τη διαδικασία έτσι ώστε να αποφανθούμε, να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, εμείς πρώτα και μετά το Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι μερικοί συνάδελφοι έχουν πολλές αμφιβολίες για την ΑΚΑ, γιατί δεν θέλουν να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Αν δείτε όμως το πρόγραμμα δράσης το οποίο εγκρίθηκε μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας του 2005 δείχνει ότι προβλέπονταν έξι, μάλλον έπρεπε να είχε εγκριθεί η συμφωνία έξι χρόνια πριν. Άρα στην ουσία θα ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο είχε αρχίσει. Δεν θα αναβαθμίσουμε τις σχέσεις μας με το Ισραήλ. Επίσης νομίζω ότι στην ουσία, εάν υπάρχει status quo στη συμφωνία, τότε αυτό θα ήταν επιβλαβές για τα δικά μας φαρμακευτικά σκευάσματα. Το Ισραήλ είναι μεγάλος εξαγωγέας ε, μεγάλων ε, ομάδων γενώσιμων προϊόντων και γι' αυτό, σύμφωνα με διάφορες μελέτες, βλέπω ότι η ΆΚΑ θα προσέδιδε προστιθέμενη αξία στα εθνικά συστήματα υγείας και τα περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι θα είχαμε ε, αποταμίευση, μάλλον θα είχαμε οικονομίες της τάξης των 100 ή 200 ε, ενός ή 2 δις ευρώ ετησίως. Και αυτό είναι ιδιαίτερα θα ήταν ιδιαίτερα ε, επικοδομητικό για μας. Ο Λάγκια ή ο Γκαντεραρίφ από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, όποιο θέλει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το θέμα επανέρχεται στην ημερήσια διάταξη. Euh, το θέμα είναι να δούμε ποια είναι η πραγματική θέση των φιλελευθέρων. Τίθεται αυτό το ερώτημα, διότι η θέση των φιλελευθέρων, τουλάχιστον όπως την εξέφρασε ε, μεγάλο διάστημα ο συντονιστής τους, ήταν να αναβληθεί η εξέταση αυτής της συμφωνίας. Κυκλοφορούν κάτι φήμες εδώ στο ράδιο Αρβίλα των Βρυξελών ότι οι φιλελεύθεροι έχουν αλλάξει θέση μετά από πίεση ιδιαίτερα του αρμοδίου επιτρόπου που είναι και δικός τους και θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση των φιλελευθέρων σήμερα. Σε περίπτωση που έχει αλλάξει, η δική μου πολιτική ομάδα θα επιθυμούσε να ακούσουμε τον Επίτροπο εδώ, τον κύριο Ντεχέχτ, στην Επιτροπή μας για να μας εξηγήσει για ποιους λόγους βιάζονται τόσο πολύ για αυτή τη συμφωνία με το Ισραήλ. Τη στιγμή ακριβώς που η κυρία Άστον στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της προσπαθεί να ασκήσει πιέσει στο Ισραήλ για να επιταχύνει τις συνευτικές διαπραγματεύσεις. Και ακριβώς στον καιρό που η Ισραηλινή κυβέρνηση δεν υποχωρεί και επιταχύνει τον επικισμό και έχω την αίσθηση, εκτός αν διάβασα λάθος, ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας ορίζεται τουλάχιστον πολιτικά, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνοχή και μια συνάφεια στις πολιτικές μας μεταξύ της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής εξωτερικών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, κάποιες αρχές και αξίες μας. Λοιπόν, αν οι φιλελεύθεροι έχουν ανακρούσει πρίμναν, θα ε, ήθελα να ακούσουμε εδώ τον Επίτροπο κύριο Ντεχούχτ να μας εξηγήσει τους λόγους, τι συμβαίνει και γιατί γίνανε αυτά, εάν η κυρία Άστον φρονεί τα ίδια και τότε θα χρειαστούμε μια ενδιάμεση έκθεση, μια προσωρινή με ε, πολιτικά και νομικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν για αυτά τα θέματα. Ε, Παρόδο, υπάρχει η κυρία Σάκα από τους φιλελεύθερους. Θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ. Χαίρομαι ότι υπάρχει αυτός ο άμεσος διάλογος και δεν κινούμεθα με φημολογίες για μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ύψης της σημασίας για μας τους φιλελεύθερους, για οποιαδήποτε χώρα και να πρόκειται και εκεί που υπάρχει παραβίαση το θέμα μας αφορά ε, άμεσα. Δεν ξέρω κατά πόσο το πρωτόκολλο είναι το κατάλληλο μέσο για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να προτείνουμε ένα χρονοδιάγραμμα μετά να προχωρήσουμε και να ψηφίσουμε. <clears throat> Well, thank you, Chairman. ο κύριος Στέρντι, συμφωνώ. Συμφωνώ με την κυρία Αντρίκενε και με τη, τους φιλελεύθερους γιατί νομίζω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτή η ομοιρία ενός τέτοιου πρωτοκόλου. Ίσως ε, ανακύψουν και νομική συμφιζητήματα, ζητήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θα πρέπει να ισχύει αυτή η εμπειρία. Όπως είπε και η κυρία Ανδρίκενε, πρόκειται για τεχνικά ζητήματα και ιατροφαρμακευτικά σκευάσματα και έχουμε να ευεργετηθούμε από αυτά. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε με αυτό το σχέδιο το ταχύτερο δυνατόν. Η κυρία Κοπά, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Όπως όλα τα θέματα που μας απασχολούν εδώ, το θέμα αυτό δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά είναι ιδιαίτερα πολιτικά φορτισμένο και σίγουρα πρόκειται για αναβάθμιση των σχέσεων μας με το Ισραήλ. Γνωρίζω ότι, όπως είπε η κυρία Αντρικέ, το θέμα αυτό είναι πλέον ε, έξι ετών, αλλά μέσα σε αυτά τα έξι χρόνια έχουν συμβεί πάρα πολλά. Και δεν έχει ε, επέλθει καμία φοβερή αλλαγή και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Συμφωνώ με τον Κατεραρίφ, είναι πάρα πολύ κρίσιμη περίοδος. Προσπαθεί η Λέδη Άστον να δώσει μια νέα πνοή ε, στις συνευτικέ συνομιλίες και για να έχουμε κάποια συνοχή και συνέπεια θα πρέπει να ε, τηρήσουμε μια στάση αναμονή, να δούμε τι θα βγει από αυτή την προσπάθεια της Λέδης Άστον και να έχουμε μια σαφή ένδειξη ότι όλα αυτά βαίνουν προς τη θετική και σωστή κατεύθυνση. Ας μην προτρέχουμε λοιπόν, ας μην βιαζόμαστε, να τηρήσουμε στάση αναμονή να δούμε τι θα βγάλει αυτή η διαδικασία. Ο Κασπάρη από το Λαϊκό Κόμμα. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Δεν έχω καταλάβει καλά, δεν είμαι βέβαιος αν κατάλαβα εντελώς αυτά που λέγουν οι συνάδελφοι. Ακούμε επικρίσεις προς τον Επίτροπο Ντεχούχτ, ότι μας έχει κάνει αυτές τις προτάσεις. Μα αυτό που έχουμε εδώ σύστημα είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κάνει τις προτάσεις και η Λέδη ε, absent, η Λέδη Απούσα και όχι Άστον, είναι μέλος των σοσιαλιστών και της σοσιαλιστικής διεθνούς. Και εκείνη είναι αρμόδια για τη συνεπή και συνεκτική κοινή εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Και πώς μπορούν οι σοσιαλιστές να το ανέχονται αυτό και να το συνδυάζουν. Ότι η συνάδελφός τους, η δική τους φέρει αυτή την απόφαση. Δεν είναι μόνο η δική μας απόφαση που έχει μπει στο αρχείο μετά τα όσα αποφασίσαμε στο Στρασβούργο για τη σχέση μας με τα Παλαιστινιακά εδάφη, όπου συμφωνήσαμε σε μεγάλη πλειοψηφία. Αλλά υπάρχει και πρόταση εδώ στην Επιτροπή μας, από την ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σταλεί από το Κοινοβούλιο, από την ίδια την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι συλλογικό όργανο η Κομισιόν για το ίδιο θέμα. Και ρωτώ ειλικρινά και ανοιχτά, γιατί οι σοσιαλιστές εδώ συνάδελφοι δεν υποστηρίζουν ε, αυτή την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υποστηρίζουν την άλλη. Και να μην καλέσουμε τον κύριο Ντεχούχτ. Κάθε φορά όποτε είχε τη δυνατότητα και τον καλούσαμε ερχόταν Αλλά τη Λέδη διάψαντα, έχω να τη δω εγώ, ξέρετε από πότε, στην Επιτροπή μας. Δεν ήρθε ποτέ. Λοιπόν, να μην καλούμε μόνο τον κύριο Ντεχούχτ, αλλά κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε να καλέσουμε και τη Λέδη Άστον, να έρθει κιόλα και να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα και με εκείνη και να μας απαντήσει και η ίδια. Γιατί δεν είναι μόνο είπατε εκπρόσωπο για την ΚΕΠΑ, διατελεί και αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μα έχει υποβάλει την ίδια συμφωνία ΑΚΑ προ ε, κύρωση. Και πραγματικά περιμένουμε πολύ μεγάλη υπομονησία τι απαντήσει που θα δώσει σε ερωτήσει ορισμένων συναδέλφων. Ο Λάγκε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κασπάρη, σωστά κατάλαβα αυτά που λέτε. Ότι συμφωνείτε να μην το προχωρήσουμε αυτό το θέμα, να μην συνεχίσουμε ε, τη διαδικασία, αλλά να καλέσουμε και τον κύριο Ντεχούχτ και την κυρία Άστον για να μας μιλήσει για τη συνέπεια της πολιτικής μας απέναντι στο Ισραήλ. Αν σας κατάλαβα καλά, συμφωνώ απολύτως με όσα είπατε. Πράγματι, να το πράξουμε αυτό, διότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου η ειρηνευτική διαδικασία ε, τρεμοσβήνει και θα πρέπει να έχουμε μια συνεπή στάση. Ωραία, να το υποστηρίξουμε. Δεν θα ορίσουμε χρονοδιάγραμμα, θα καλέσουμε τους δύο επιτρόπους και να συζητήσουμε εδώ για τη συνέπειά μας ε, στην πολιτική μας απέναντι στο Ισραήλ. Καντέρα Ρίφ. Λατρεύω τον Ντανιέλ Κασπαρί φαίνεται ότι υπερασπιζόμαστε τον Ντεγκούχτ, μάλλον ή αντιτιθέμεθα, υποστηρίζοντας τη Λέδη Άστον. Μα μας, μας ενδιαφέρει η ουσία. Εάν συμφωνείς, εντάξει, μπορούμε να ακούσουμε και τον με και την δε. Και αν δεν συμφωνούμε με τη Λέδη Άστον, θα πούμε, παρόλο που είμαστε σοσιαλιστές, θα το πούμε. Δηλαδή δεν προστατεύουμε την οικογένειά μας υπό τη στενή έννοια. Ο συνάδελφος το έθιξε. Εάν συμφωνούμε και πούμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και να δούμε ποια είναι η θέση της Κομισιόν μέσω των δύο επιτρόπων, ας δούμε κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε σε μια πολιτική συνένεση και μετά να προβούμε σε μια ακρόαση, να προχωρήσουμε σε μια ακρόαση έτσι ώστε να δούμε επί της ουσίας τι, σκεφτούμε, τι σκεφτόμαστε επί του θέματος. Συμφωνώ με τον Μπέρντ. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να συζητάμε και τα θέματα αυτά φτάνοντας σε μία σύμπνοια, Ντανιέλ. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία συγκεκριμένη πρόταση. Θα δώσω το λόγο σε όλους. Τέσσερις ζητούν το λόγο. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τις σκεφτόσαστε ως προς την ε, πρόταση Κανταρεΐφ. Πριν προχωρήσουμε και ακούσουμε τον Επίτροπο Ντεχούχτ και την Επίτροπο Άστον. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη πρόταση. Τι τι σκέφτεστε επ' αυτής της πρότασης, να ακούσουμε τους ε, δύο επιτρόπους, Ντανιέλ Κασπαρή. Ναι. Προσοχή για να συνεννοούμαστε και να μην διαστρεβλώνουμε αυτά που λέμε, καμιά φορά και στην ίδια γλώσσα. Εδώ μιλούμε για κοινή εξωτερική πολιτική ε, και τη συνέπειά της ε, προς ε, τους εταίρους μας. Αυτό δεν το αμφισβητεί το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εσείς το αμφισβητείτε, οι σοσιαλιστές, που είπατε ότι χρειάζεστε να συζητήσετε με τον Τεχέχτ και την Άστον για αυτό το θέμα. Εγώ να δείτε σε πόσα θέματα θέλω να συζητήσω μαζί τους. Αλλά όχι γι' αυτό το θέμα της συμφωνίας ΑΚΑ με το Ισραήλ. Έχει κάνει τόσες προτάσεις και τα θέματα της Αλίας και της Γεωργίας με τους Παλαιστινίους τα έχουμε διεκπαιρεώσει και αυτό το άλλο θέμα είναι από την ίδια Επιτροπή και από την ίδια ύπατη εκπρόσωπο που διατελεί κατά τα άλλα όπως σας είπα και αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το έχουμε κάνει τεράστιο ζήτημα αυτό. Δεν κατάλαβα. Δεν θα πρέπει να... Ε, έχουμε ομήρου τώρα με μονομένα θέματα. Αν θέλετε να συζητήσουμε για τη συνέπεια τη εξωτερική πολιτική, δεν θα διαχωρίζουμε τα θέματα. Η πολιτική εξωτερικών υποθέσεων θα πρέπει να μας στείλει τη γνωμοδότησή τη για αυτό το θέμα, τη Συμφωνία ΣΑΚΑ και ε, ε, θα διαμορφώσουμε άποψη για ανεξάρτητα από αυτό Τελείω ανεξάρτητα υποστηρίζω την πρόταση να καλέσουμε και τον κύριο Ντεχούχτ και τη Λέδη Άστον ε, στην Επιτροπή μα και να του ακούσουμε. Γιατί πραγματικά αυτό το θέμα τη συνέπεια και συνοχής της ε, πολιτική εξωτερικού και διεθνού εμπορίου συνδέεται με την εξωτερική πολιτική. Και δεν είναι μόνο θέμα Ισραήλ και Παλαιστινιακών εδαφών, είναι μια σειρά άλλα θέματα που μας απασχολούν εδώ, πολλά και διάφορα. Thank you. Κύριε Σόλτς, ευχαριστώ πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να έχουμε πολιτική συνέπεια αλλά είναι η συνέπεια της πολιτικής και όχι συνέπεια μεταξύ διαφόρων χαρτοφυλακίων, διαφόρων επιτρόπων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μια πολιτική διαδικασία πολύ ευαίσθητη και λεπτή και η θέση της σοσιαλιστικής ομάδας στην Επιτροπή μας εδώ είναι πάρα πολύ λογική και πάρα πολύ σωστή και πάγια. Θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση επιτόπου συγκεκριμένα. Δεν πρόκειται για διάφορα παιχνιδάκια μεταξύ πολιτικών ομάδων, είμαστε υπέρ κατά ενός επιτρόπου. Το θέμα είναι να έχει μια υπεύθυνη στάση η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο, σε μια πάρα πολύ εύθραυστη και ευαίσθητη περιοχή του κόσμου. Και όχι απλώς τρεμοσβήνει ε, η διαδικασία όπως είπε ο κύριος Λάγκε. Ποια διαδικασία ειρηνευτική, εγώ δεν τη βλέπω καν να τρεμοσβήνει, είναι σβηστή. Ναι, λοιπόν, στην πολιτική συνέπεια και στη συνέπεια της πολιτικής μας να γίνει συζήτηση. Θα φέρουμε όμως τρεις επιτρόπους, παρακαλώ. Θυμίζω ότι και ο Επίτροπος Φούλε είναι αρμόδιος γιατί συζητάει για θέματα νότιας γειτονίας και τα έχει και αυτά τα θέματα υπόψη του και τα χειρίζεται. Λοιπόν, να καλέσουμε τρεις επιτρόπους. Την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δύο επιτρόπους για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να καταλάβουμε τι πολιτική θέλουν να ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με τις χώρες αυτής της περιοχής. Ευχαριστώ. Thank Robert Πρόεδρε, μου φαίνεται ότι θα ζητήσουμε όλο το κοινοβούλιο τελικά και θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει τελικά και την έκθεση. Αν θέλετε να ακολουθήσετε την λογική της κυρία Σκοπά, η έκθεση της δεν θα είχε περάσει το κοινοβούλιο και εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, διότι ε, ε, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχω περί κάποια πλευρά, ούτε προ τη μια ούτε προ την άλλη πλευρά. Ε, όμως ήδη παίρνουμε το, μέρος, το, το ένα μέρο ή το άλλο μέρο. Ε, ένα μέρο υποστηρίζει τη μια πλευρά και άλλο την άλλη. Πιστεύω ε, ότι ε, αφού περάσαμε την ομάδα ε, Γεωργιάς και Αλίας για τους Παλαιστινίους, θα πρέπει να ακολουθήσουμε και αυτό. Μπορεί να απορριφθεί, αλλά ας δώσουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε. Όσο πιο πολλοί συμμετέχουν, τόσο πιο πολύ θολώνουν τα νερά στο τέλος. κυρία, Σάκα. Ναι, ποιος μπορεί να ενταχθεί σε μια τόσο υπέροχη λίστα ατόμων που μπορούν να μας επισκεφθούν και να συζητήσουμε για νέες πολιτικές στον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να είμαστε ειλικρινεί και να δούμε τι αποτελεί τεχνική και τι αποτελεί πολιτική συζήτηση. Όλοι γνωρίζουμε τις τάσεις που διακυβεύονται και είναι σημαντικό για τη δική μας αξιοπιστία, για τη δική μας συνέπεια να ε, δούμε τα θέματα στην ουσία τους. Και βέβαια αυτό είναι πολύ ευαίσθητο, είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα αυτά, αλλά ας κοιτάξουμε και τη δική μας θέση εδώ ο κύριος Αρίφ, θα πρέπει να αποφύγουμε κάτι εδώ. Θα πρέπει να μην ε, πιστεύουμε ότι έχουμε διαλέξει να πάρουμε το μέρος ενός στρατοπέδου εναντίον Δεν είμαι υπέρ κάτι ή κατά κάποιο άλλου θέματος, διότι μετά μπαίνουμε σε πολύ περίπλοκα ε, πολιτικά και ευαίσθητα θέματα. Και ε, δεν θα ήθελα να το κάνουμε αυτό, διότι θα ήταν πολύ επικίνδυνο για μας να το δούμε από αυτή την οπτική γωνία. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πούμε αυτό το θέμα έχει αναφερθεί και από άλλους, δεν είναι τεχνικό ζήτημα. Όταν βλέπουμε τη συζήτηση για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, την, τις πιέσεις που γίνονται από πλευράς Αμερικής για να μην αναγνωριστεί, τις σχέσεις ε, που υπάρχουν και μετά όλα τα πολιτικά ε, κόμματα σε Ευρωπαϊκή ε, Ένωση όπου βλέπουμε την Ευρώπη να συμμετέχει σε αυτή την ηνευτική διαδικασία ε, περισσότερο. Και εγώ είμαι για μια ισχυρή πολιτική Ευρώπη για να έχει το βάρος της σε αυτό το μέρος της Ιφιλίου. Βέβαια, εδώ αναρωτιόμαστε. Δεν είναι τεχνικό, τεχνική πράξη, είναι πολιτική πράξη. Εγώ δεν ζητάω τίποτα περισσότερο. Είναι να πούμε, να εξετάσουμε και να δούμε με όλα τα στοιχεία, να έχουμε τη δυνατότητα και η μεν και η δε, να πούμε ποια είναι τα ερωτήματά μας, οι αμφιβολίες μας κλπ. Και να ε, έχουμε εδώ να υποδεχτούμε τους τρεις επιτρόπους γιατί αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, να εκφραστούν διάφορα θέματα και θα δούμε σε εκείνη τη φάση πώς μπορεί να προχωρήσει στην ουσία αυτός ο φάκελος. Ε, πέρα από τις πιέσεις και τα άλλα που μπορεί να υπάρχουν, εγώ ε, δεν ζητάω τίποτε παραπάνω, δεν θέλω να ε, δημιουργηθούν αυτές οι διαδικασίες έντασης ανάμεσά μας. So, we have Διαδικαστικό ζήτημα πριν μπούμε στο ουσιαστικό. Τι να κάνουμε τώρα, πώς θα συνεχίσουμε. Προτείνει ο Καντέρα Ρίφ πριν προχωρήσουμε να καλέσουμε τρεις επιτρόπους. Φτάσαμε στους τρεις, έτσι. Ωραία. για να έχουμε μια συνολική εικόνα του θέματος. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε πρώτα για αυτό το διαδικαστικό ζήτημα. Εντάξει, συμφωνείτε. Ποιοι είναι υπέρ αυτού του διαδικαστικού αιτήματος. Διαδικαστικό είναι. Λοιπόν, τι ακριβώς προτείνετε κύριε Κασπάρη. Προτείνω, όπως πάντα είτε να ψηφίσουμε, οπότε θα ψηφιστεί στη ώρα των ψηφοφοριών, είτε μιλάμε για διαδικασία και αυτό θα το λύσουν οι συντονιστές. Ναι, έχετε δίκιο. Τα διαδικαστικά ζητήματα τα λύνουν οι συντονιστές κανονικά κατά τη διάρκεια της δικής του συνεδρίασης. Οπότε τα αφήνουμε όπως έχει. Υπάρχει συγκεκριμένη πρόταση για τη διαδικασία για το θέμα ουσίας τώρα. Προς το παρόν δύο είναι οι θέσεις, αν κατάλαβα καλά. Η μία είναι να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη και η άλλη είναι να μην δώσουμε, να την αναβάλουμε, όχι να απορρίψουμε. Ε, κανείς δεν έχει προτείνει απόρριψη της συμφωνίας ακόμα. Απλώς να αναβάλουμε την ε, χορήγηση της σύμφωνης γνώμης. Ο Κασπάρη. Ναι, αγαπητέ Πρόεδρε. Ζήτησα η ΑΦΕΤ, η Επιτροπή Εξωτερικών, να μας στείλει τη γνωμοδότησή της, γιατί θέλω να αποφασίσω και να δω τι λέει η Επιτροπή Εξωτερικών για αυτό το θέμα. Γιατί υπάρχουν και άλλα πιο σημαντικά θέματα από τα εμπορικά. Ναι, ναι, βεβαίως. Η ΑΦΕΤ περιμένει εμά λέει ο πρόεδρος, να στείλουμε χρονοδιάγραμμα. Και εμεί περιμένουμε εκείνου να στείλουν γνωμοδότηση. Κυρίες και κύριοι, θα διαβιβάσω στην Επιτροπή Εξωτερικών το αίτημά σας να προχωρήσουν ε, στη γνωμοδότησή τους και θα δούμε τι θα αποφασίσουν για τα διαδικαστικά στη συνέχεια οι συντονιστές και θα φέρουμε χρονοδιάγραμμα για όλο το θέμα. Εντάξει, συμφωνήσαμε. Ωραία. Let's move to... Προχωρούμε. Σημείο 6. η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ουσμπεκιστάν. Επέκταση των διατάξεων της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας στο διμερές εμπόριο εφαντουργικών προϊόντων. Είναι η τρίτη φορά που ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Πρόκειται για ένα σχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης, δεύτερη εξέταση, διότι έχει συζητηθεί ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση. Η συγητή μα είναι ο Τζορτ Σάπιν Κούτα, Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε, και θα του δώσω μέσα το λόγο. Προηγουμένω, θα ήθελα να σα πω ότι. Ο πρέσβης του Ουσπεκιστάν αποφάσισε να μην δεχτεί τις επανειλημμένες μας ε, προσκλήσεις να έρθει στην Επιτροπή. Μου, μου απίφθινε ε, ε, επιστολή και μου είπε ότι θέλει να έρθει η πρέσβης αλλά να μην τις κάνουμε ερωτήσεις. Ε, μάλλον στην αρχή είπε θα έρθει ο πρέσβης, αλλά να μην κάνουμε ερωτήσεις. Μετά είπε να στείλει κάποιον άλλον. Εγώ είπα όχι, δεν μπορούμε να δεχόμαστε τέτοιου όρου όταν καλούμε ένα πρέσβη, καλούμε πρέσβη να συμμετέχει ε, στην Επιτροπή μα και συζήτηση. Και του είπα να μου στείλει γραπτή δήλωση, ε, αν θέλει να την αναγνώσουμε. Έστειλε λοιπόν μια γραπτή δήλωση, κυκλοφόρησε και τώρα επισήμως η θέση ε, των Ουσμπέκων ε, και της εδώ αποστολή τους ε, είναι γνωστή και γραπτός διατυπωμένη. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον εισηγητή μας πρώτα, τον κύριο Κούτας και βλέπουμε. Uh, thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Πρέπει να πω ότι λυπάμαι που δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τον πρέσβη. Είναι η τρίτη φορά που πεθύνουμε την πρόσκληση, δυστυχώς και προφανώς ε, ε, δεν επιθυμεί να έχει αυτό το διάλογο μαζί μας. έχετε την άποψή τους, την έχουμε διανύμει, την έχετε μπροστά σας. Θα πρέπει να πω ότι είχα και την ευκαιρία να συναντηθώ εγώ προσωπικά με τον ε, Περέσβη. Προσπάθησε να μου εξηγήσει την κατάσταση ε, λίγο πολύ γιατί το Ουσβεκιστάν δεν πολύ βαμβάκι ε, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ε, προϊόντων πια. Και όταν ήγερα το θέμα μιας ανεξάρτητης αποστολής ε, του ΔΟΕ στο Ουσμπεκιστάν, η απάντηση ήταν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την έκθεση της UNICEF. Της UNICEF είναι ο μόνος διεθνής οργανισμός που έχει παρουσία στο Ουσβεκιστάν αυτή τη στιγμή. Επίσης, ε, ε, βλέπω την παρουσία, την παρουσία της UNICEF θετική, αλλά δεν μπορεί να υποκαθιστά ε, τη λειτουργία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ως οργανισμός παρακολούθησης. Επίσης, συμμετείχα σε μια συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και οργανώθηκε από την ΑΦΕΤ όπου εκπροσωπήθηκε και η UNICEF και παρουσίασε τη θέση της σχετικά με το Ουσβεκιστάν και είπαν ότι παρόλο που παρατήρησαν ότι έγιναν θετικές αλλαγές ε, υπάρχει ακόμη πολλής δρόμος ε, να διανύσουμε στο τομέα της παιδικής εργασίας. Αυτή είναι και η θέση της UNICEF λοιπόν. Στο μεταξύ Μόλις έλαβα και τη γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής Εξωτερικών ε, και την προσωρινή έκθεση και πρέπει να σας πω ότι ε, υπάρχει συντριπτική πλειοψηφία. Όλοι υπερψήφισαν αυτή την προσωρινή έκθεση. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αν θέλουμε να ξέρουμε μια λύση θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, είναι καλό να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν, διότι έχουν ε, συναντηθεί με τον πρέσβη, αλλά για μένα είναι σαφές ότι ε, όπως έχουν τα πράγματα δεν μπορούμε να έχουμε αυτόν τον διάλογο με την πλευρά των Ουσβέκων. Ε, έχουμε τον κύριο Φιλίππ Κισόν από πλευρά της Κομισιόν και δίνω το λόγο κατευθείαν τον ε, πρόσωπο της Κομισιόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα θυμάστε όταν είχαμε συζητήσει τα τέλη Αυγούστου αυτό το θέμα την προηγούμενη φορά, είχαμε πει ότι θα είχαμε συνάντηση με τον πρέσβη του Ουσβεκιστάν στι 7 Σεπτεμβρίου και αυτή η συνάντηση ήταν στα πλαίσια των προσπαθειών που είχαμε καταβάλει για τη διάσκεψη τη ΔΟΕ για να επιταχύνουμε τις διπλωματικές προσπάθειες με το Ουσβεκιστάν. Σε εκείνη τη συνάντηση επιμείναμε κυρίω σε δύο ζητήματα. Πρώτον, και πιστεύω ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το ακούσουμε αυτό είχαμε πει στον Πρέσβη ότι έπρεπε να ξεκινήσει ένα διάλογο με την Επιτροπή ΙΝΤΑ στο θέμα της παιδικής εργασίας. Κατά δεύτερο λόγο, οθήσαμε το Ουσβεκιστάν με ε, πολύ ε, σεναρούς όρους να υποδεχτούν, να δεχτούν την πραγματοποίηση μιας αποστολής της ΔΕΣ στο Ουσβεκιστάν ε, Ε, λυπούμαστε που δεν ήταν δυνατό να έχετε αυτή τη συζήτηση σήμερα με τον πρέσβη σε αυτή την Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την αποστολή της ε, ΔΟΕ, ε, το Ουσμπεκιστάν ε, άκουσε το μήνυμά μας σχετικά με την σημασία που είχε αυτή η αποστολή και πιστεύουμε ότι μεταδόθηκε από τον πρέσβη το μήνυμα αυτό στις αρχές του Ουσμπεκιστάν και ότι εξετάζεται το θέμα. Η πλευρά ε, του Ουσμπεκιστάν αυτή τη στιγμή είπαν ότι ε, συζητούν με την ΔΟΕ. Το περασμένο Αύγουστο έδωσαν ε, μία έκθεση για την υλοποίηση της σύμβασης εργασίας η ΔΟΕ που επισημερινευάνει και την παιδική εργασία σύμφωνα με τους κανόνες της ΔΟΕ. Επίσης έδωσαν πληροφορίες σχετικά με ένα σχέδιο δράση το οποίο είχε εγκριθεί το Σεπτέμβριο με στόχο την διασφάλιση της σωστής υλοποίησης της σύμβασης της ΔΟΕ. Η πλευρά των επίσης υπογράμμισε ότι η συνεργασία με την UNICEF δείχνει ότι, δεν, ε, ότι δείχνουν κάποια συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς και έχουν τονίσει ότι θα δώσουν ε, βοήθεια στην, στα γραφεία της UNICEF που ε, διενεργεί εργασίες παρατήρησης και παρακολούθησης στην, κατά διάρκεια της συλλογής του βαμβακιού από τα παιδιά. και παράλληλα η Κομισιόν θα παρακολουθεί από ε, κοντά τις εξελίξεις στην φετινή συλλογή του Παπακιού με την βοήθεια πληροφοριών από μια νέα προσωπία που έχουμε εκεί και από τις πρεσβείες των κρατών μελών. Ε, οι πρώτες ενδείξεις ε, δείχνουν ότι υπάρχουν κάποιες ε, βελτιώσεις αλλά θα πρέπει να παραμείνουμε θα περιμένουμε μέχρι να δούμε το τέλος της διαδικασίας συγκομιδής. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η αποστολή της ΔΟΕ στην Ουσπεκιστάν είναι το κλειδί για τη διασφάλιση μιας βελτίωσης της κατάστασης του Ουσπεκιστάν. Άρα θέλουμε να επιταχύνουμε επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας για να πείσουμε τις ε, αρχές του Μεκιστάν να αποδεχτούν την πραγματοποίηση μιας τέτοιας αποστολής από την ΕΔΟΕ. Αν η ΔΟΕ θεωρεί ότι είναι ε, ε, ότι θα βοηθούσε. Είμαστε έτοιμοι εμείς να στείλουμε μια ομάδα στη Σασκένδη μέχρι τα τέλη του Οκτώβρη, για παράδειγμα. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι πιστεύουμε ότι είναι θετικό και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν να αξιολογήσουν την κατάσταση στο Ουσμπεκιστάν και να δώσουν ε, την δυνατότητα στους Μπέκους να λάβουν θετικά μέτρα. Αυτό συνάδει με την προσέγγισή μας σχετικά με την παιδική εργασία και την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και να δούμε τους λόγους για τους οποίους πρώτα απ' όλα τα παιδιά δουλεύουν στους αγρούς, όπως για παράδειγμα την έλλειψη της ε, χρήσης μηχανημάτων στην γεωργία στο Οσμπεκιστάν. Θα σας αναφέρουμε ε, όταν υπάρχουν οποιασδήποτε εξέλιξεις. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ χρήσιμες οι πληροφορίες αυτές. Ας πάμε στα άλλα μέλη της Επιτροπής. κύριε Κόπα. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή ΑΦΕΤ έχει στείλει ένα πολύ στεναρό ε, μήνυμα στην κυβέρνηση του Ουσμπεκιστάν λέγοντας ότι δεν αποδεχόμαστε δηλώσεις εκ μέρους της κυβέρνησης πια. Θέλουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ε, για την Επιτροπή ΑΦΕΤ η ε, αποστολή παρακολούθησης της ΔΟΕ θα πρέπει να συνεχίσει χωρίς οποιαδήποτε συμφωνίες ή αναβαθμίσεις συμφωνιών. Όχι μόνο να υπάρξει αυτή η αποστολή αλλά να έχουμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα που να δείχνουν αλλαγή προσανατολισμού και θέσεις ό,τι αφορά την παιδική εργασία. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πραγματικά ότι ζητήματα όπως η παιδική εργασία αποτελούν δοκιμασίες για μας ε, για να δούμε αν πραγματικά τηρούμε τις αξίες μας. Και συμφωνώ με τον εισηγητή και την ε, Κομισιό ότι προτού λάβουμε οποιασδήποτε συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά του Ουσβεκιστάν ε, να μην προχωρήσουμε. Ο Πολ Μέρφυ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή. Κρίμα που δεν έχουμε εδώ εκπρόσωπο του πρέσβη, της πρεσβείας. Είναι ενδεικτικό ε, για τη στάση τους, όπως και ο πρόεδρος. Έχουμε ένα σημείωμα και βασικά αυτό που λένε ε, είναι ότι δεν, δεν τηρούν τις ε, διατάξεις ε, ούτε κυρώνουν τις συμφωνίες. Μπορεί να έχουν κυρώσει στη θεωρία της συμφωνίας του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, αλλά στην πράξη δεν το υλοποιούν. Ευχαριστώ που μας ε, ενημερώνετε. Ξέρετε ότι εκεί όλοι οι Γεωργία λένε, ακόμα και η συλλογή του βαμβακιού είναι στα χέρια των ιδιωτών αλλά έχουν ε, ημερήσια ποσόστοση που θα πρέπει και το επιβάλλει το κράτος. Και αν κάποιος δεν ε, θέλει να δουλέψει, δεν μπορεί να δουλέψει, πρέπει να έχει χρήματα για να πληρώσει κάποιον άλλο στη θέση του, να πάει να μαζέψει ε, τη ποσόστοση της ημέρας. Και πάλι, και τώρα είναι η περίοδος ε, της ε, συγκομιδής. Ένας φοιτητής έστειλε ένα γράμμα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και ζητάει βοήθεια. Μας βασανίζουν με τρόπο φασιστικό, μας πηγαίνουν ε, στις φοιτίες 4 η ώρα το πρωί, πρέπει να μαζεύουμε 100 κιλά τη μέρα, δεν έχουμε νερό και διαμαρτυρήθηκε και ζήτησε το λόγο από ένα δάσκαλο και ο δάσκαλος το αντέκρουσε και είπε ότι τα παιδιά πηγαίνουν ε, στις 7 η ώρα στα χωράφια σηκώνονται 5, 5,5 ώρα ή 6 πηγαίνουν με τη βούλησή τους γιατί τους αρέσει και ε, κοιμούνται στις 10 η ώρα και μαζεύουν 5 κιλά βαμβάκι αυτά λέει η άλλη πλευρά η δάσκαλη είναι καταναγκαστική παιδική εργασία και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συνεχίζεται στο Ουσμπεκιστάν. Πραγματικά χρειάζεται ανεξάρτητη ε, επιβεβαίωση ε, αυτής της κατάστασης για να προχωρήσουμε. Ο Ντανιέλ Κασπάρη από το ΕΛ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κατά την άποψή μου πρέπει να σας πω ότι έχω καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από το ψήφισμα της Επιτροπής Εξωτερικών θέλω να τονίσω τα σημεία 5 και 8 που ε, γίνονται πολύ ρητές αναφορές για το πού θα υπάρξουν βελτιώσεις και πού χρειάζονται βελτιώσεις. Βεβαίως θα πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα και συμφωνούμε ότι δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη. Ούτε θα έχουμε αύριο ανθυρά τοπία και την κατάσταση όπως ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω καλό είναι να διατηρήσουμε κάποια πίεση και θεωρώ ότι η Ουσμπεκική πλευρά γνωρίζει και καλό είναι να γνωρίζει ε, τι μηνύματα θα πρέπει να μα δώσει και χειροπιαστές ε, αποδείξεις. Ε, θα ήμουν ευγνώμων αν ο εισηγητή μα έκανε μια πρόταση προ την κατεύθυνση αυτή μέχρι που θα συμπεριλάβει στην έκθεσή του τα όσα συμπληρώσει η Επιτροπή Εξωτερικών και είμαι βέβαιος ότι και εδώ στην Επιτροπή μας θα υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία για την έκθεσή του. Uh, Από το Alde η Κατρίν Μπίρντε. Θα ήθελα να πω ότι στην τελευταία μας συνάντηση τάχθηκα υπέρ του να παρευρεθεί εδώ ο πρέσβης και θεώρησα ότι θα πρέπει να του δώσουμε μια ευκαιρία να μας μιλήσει. Αποφάσισε να μην το κάνει και μας έστειλε μια γραπτή απάντηση. Και στο τέλος σελίδας 1 αναφέρεται ότι η, ε, ελάχιστη, η, η κατώτερη ηλικία απασχόλησης είναι τα 16 χρόνια. Και άρα έχουμε ε, σαφή στοιχεία ότι κάτι τέτοιο έχει παραβιαστεί, η συμφωνία είχε παραβιαστεί σε σχέση με αυτούς που συμμετέχουν στη συγκομιδή, εκείνους που οδηγούν τα παιδιά ε, στο, στις καλλιέργειες, στα σημεία συγκομιδής και νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δεν διαθέτουμε πλέον άλλη υπομονή, θα πρέπει να τους παραπέμψουμε. Βρισκόμαστε σε φάση συγκομιδής και αν το αφήσουμε τώρα θα περάσει ένας κύκλος ε, πάλι εμπορίας, συγκομιδής και εμπορίας πριν ξανασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Ήμασταν αρκετά ανεκτικοί, προσπαθήσαμε να τους δώσουμε αρκετές ευκαιρίες, ήμασταν δίκαιοι υπέρ το οδέων. αλλά νομίζω ε, ότι ε, δεν μας φέρονται σωστά, είναι ιδιαίτερα θρασής απέναντί μας και δεν μπορούμε να το δεχτούμε πλέον αυτό. Ευχαριστώ τους συναδέλφους, όλους τους συναδέλφους για τις θέσεις σας στην έκθεση για να απαντήσω στον κύριο Κασπάρη, θα ήθελα να λάβω υπόψη όλες τις γνωμοδοτήσεις, αλλά η προθεσμία είναι Παρασκευή για την υποβολή τροπολογιών. Μπορείτε να υποβάλλετε οποιασδήποτε τροπολογίες επιθυμείτε εγώ είμαι έτοιμος να τη συζητήσω και να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό γιατί θα ήταν σκόπιμο να έχουμε μια ιδιαίτερα ισορροπημένη έκθεση. Εγώ κρατάω θετική στάση. Είμαι υπέρ του καρότου και όχι του μαστιγίου γενικά. Αλλά μερικές φορές όταν δεν μπορεί να γίνει διάλογος τι να κάνουμε, ραβδοκοπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει συμφωνία λοιπόν επί του θέματος και από πλευράς Επιτροπής ε, η υποβολή τροπολογιών μέχρι τις 14 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε την έκθεση στις 22 Νοεμβρίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος συνεχίζει χωρίς μικρόφωνο. Περνάμε στο θέμα 7 και πάλι χωρίς μικρόφωνο. Ο Πρόεδρος, ε, Σύστημα Γενικευμένων δεσμολογικών Προτιμήσεων. Ο, κυρ, ο Κρίστοφερ Φιέλνερ από το ΕΛΚ, ο εισηγητής, έχει υποβάλει ένα έγγραφο εργασίας το οποίο έχετε στη διάθεσή σας. Άρα Θα συζητήσουμε αυτό το εγγραφό. Δίνω το λόγο στον κύριο Φιέλνερ. για να σχολιάσει το έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνουμε το εξής. Δεν θα ήθελα να δούμε λεπτομεριακά το έγγραφο, γιατί ξέρω ότι οι συνάδελφοι αφιέρωσαν χρόνο για να διαβάσουν το κείμενο αυτό και γι' αυτό δεν θα ήθελα να σας εξαναγκάσω να τα ακούσετε για άλλη μια φορά. Θα ήθελα εντάχει να πω ότι σε αυτό το έγγραφο εργασίας προσπάθησα να κατακαιρματίσω την πρόταση σε διάφορες συστάδες. Να δούμε δηλαδή πού θα πρέπει να κινηθούμε για να αποφασίσουμε. Η πρόταση της Επιτροπής είναι καταρχήν καλή, αλλά θα πρέπει να δούμε τι πρέπει να αλλάξει. Αφού αναφερθώ σε αυτές τις επιμέρους συνιστώσεις, θα ήθελα να ακούσω απόψεις, να μου πείτε δηλαδή εάν θα πρέπει να μας απασχολήσει κάτι ιδιαίτερα. Νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι αυτό το έγγραφο βάση συζητήσεων. Η πρώτη συνιστός είναι η γεωγραφική κάλυψη. Μπορούμε να δούμε πόσες χώρες υπάρχουν, πόσες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν. Εμείς θα πρέπει να συμφωνήσουμε ποια θα πρέπει να είναι η συστηματική μας προσέγγιση. Όπως ξέρετε στην πρόταση αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το μέσο εισόδημα που ορίζει η Παγκόσμια Τράπεζα για τις χώρες αυτές και θα ήθελα τα σχόλιά σας. Τι σκέφτεστε επί του θέματος. Έχει σημασία να έχουμε προβλέψιμα μέσα. Ως προς την κάλυψη προϊόντων, η Επιτροπή δεν αλλάζει την κάλυψη προϊόντων. Εμείς θα πρέπει να αποφασίσουμε κατά πώς θα πρέπει να μας απασχολήσει και η κάλυψη προϊόντων, διότι με την πρόταση της Κομισιόν αποκλείονται αρκετές χώρες και θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα ευαίσθητα και μη προϊόντα δυνάμει του κανονισμού αυτού. Η δεύτερη δέσμη αφορά τη διαβάθμιση και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα χρησιμοποιήσουμε το GSP Plus, δηλαδή το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν και κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχουν κατόφλια στη διαβάθμιση αυτή, μέσα στα πλαίσια αυτής της ε, διαβάθμισης. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να προσαρμοστεί το όλο πλαίσιο με όλες αυτές τις χώρες οι οποίες αποκλίνονται. Θα πρέπει να αποφασίσουμε και να δούμε κατά πόσο είναι σωστό ή εσφαλμένο αυτό και να δούμε κατά πόσο αυτά τα νέα αριθμητικά στοιχεία ε, οδηγούν σε μία αντιστήχηση με την με τις χώρες που περιλαμβάνουμε. Ως προς το, την ε, τρίτη, την τέταρτη συνιστόσα είναι το GSP-SYN, δηλαδή οι επαυξημένες δασμολογικές προτιμήσεις και κατά πόσο θα είχαμε δύο νέες χώρες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το μηχανισμό GSP GSP-SYN+. Νομίζω ότι θα πρέπει το GSP Syn plus να γίνει δελεαστικό. Γιατί απλουστεύοντας ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων ισχύει γιατί εμείς είμαστε οι ευεργέτες. Το GSP Plus όμως είναι κάτι γιατί υπάρχουν ευεργετήματα και για εμάς. Υπάρχουν ευεργετήματα για όλο τον κόσμο. Άρα οι χώρες που πληρούν αυτές τις προδιαγραφές και που δέχονται αυτή τη συμφωνία θα έχουν ακόμα πιο προτιμησιακές συμφωνίες μέσα στα πλαίσια των εμπορικών συναλλαγών. Αλλά το GSP Plus θα πρέπει να γίνει ακόμα πιο προτιμησιακό, δηλαδή πιο δελεαστικό. Και είναι πράγματι σε σχέση με το GSP με το αρχικό σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά είναι αρκετά προτιμησιακό. Δεν είναι. Δίνει ευεργετήματα για αυτές τις χώρες. Για τις χώρες όπου υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές ως προς τη διακυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής. Αλλιώς ποια είναι η αξία του GSP+. Όπως είπα εξ αρχής, δεν θα με ε, ενδιέφερε να αλλάξω αυτό τον κατάλογο των 27. Ε, εάν αρχίσουμε με αυτή την άσκηση, δεν ξέρω ποιες από τις 27 ή 30 συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι η συμφωνία είναι βάσιμη και δεν θα ήθελα να αλλάξει κάτι. Υπάρχει μια σύμβαση που δεν έχουμε κυρώσει εμείς, η Σουηδοί. Η Σουηδία δεν την έχει κυρώσει, η χώρα μου δηλαδή. Πάση περιπτώσει δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δελεαστικό αυτό το σύστημα, το σύστημα ΣΥΝ ή όχι. Αφήνω το 5 και πάω στο 6, δηλαδή στις ρήτρες διασφάλισης. Ό,τι και να κάνουμε, θα πρέπει να έχουμε επαρκείς διασφαλίσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Και η Επίτροπη έχει ενισχύσει τις ρήτρες διασφάλισης. Αρκούν. Είναι επαρκείς. Χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Αφήνω το 7 τη διαδικασία επιτροπολογίας. Την αφήνω κατά μέρο, ευπρόσδεκτα βεβαίω τα σχόλια από τη δική σας πλευρά ως προς το 8, την διάρκεια ισχύω του κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να ισχύει στο δινεκές, δηλαδή να είναι αορίστου χρόνου του χρόνου δεν, δεν μου έχει καλό. Ίσως θα πρέπει να μπορούμε να, να θεωρήσουμε κάποια στιγμή τη στιγμή που θα επέλθουν και ουσιώδεις αλλαγές. Θα ήθελα όμως και τη δική σας άποψη. Λοιπόν, γεωγραφική κάλυψη, κάλυψη προϊόντων, διαβάθμιση, GSP-SYN, RIT ρήτρες διασφάλισης και διάρκεια. Αυτές είναι οι βασικές συνιστώσεις επί των οποίων θα πρέπει να αποφασίσουμε. Εδώ θα ήθελα να μου πούν και οι συνάδελφοι τι σκέφτονται, τι πρέπει να κάνουμε στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει και ο Πρόεδρος. Τα έγγραφα εργασίας είναι πολύ χρήσιμα. Μπορούν να σταθούν πολύ χρήσιμα. και να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για συζήτηση. Ο Ρόμπερτ Στέρντι από τη, τους Ευρωπαίους μεταρρυθμιστές και συντηρητικούς. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Κρίστοφερ και θα ήθελα να συγχαρώ την Κομισιόν γιατί δεν ήταν εύκολο το έργο της Κομισιόν για να αποφασίσει ποιες χώρες συμπεριλαμβάνονται και ποιε όχι, διότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι μια-δυο χώρε ας πούμε, θα έπρεπε να παραμείνουν και άλλες θα έπρεπε να βγουν. Εάν όμως ακολουθούσαμε αυτό το δρόμο δεν θα φτάναμε σε κάποια επίλυση του ζητήματος. Ως προς την διαβάθμιση Νομίζω ότι ευεργετεί πλούσιες χώρες όπως τις είπα και την Ελβετία. Και αυτό με απασχολεί πραγματικά για τον τρόπο διαβάθμισης που έχετε ορίσει. Δηλαδή, η Κομισιόν θεωρούσε ότι οι χώρες μεσαίου εισοδήματος δεν θα πληγούν με βάση αυτό το σύστημα διαβάθμισης, αλλά θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία παγιοποίηση των προτιμήσεων, των προτιμησιακών συμφωνιών που ήδη προϋπάρχουν. Θα ήθελα να υποβάλω την εξής ευθύτατη ερώτηση προς την Επιτροπή. Εγώ πάντα συμμετείχα στην ΙΤΑ και θεωρώ το εμπόριο είναι καλύτερο από την αρρωγή. Γι' αυτό πιστεύω στις προτιμησιακές, στις γενικευμένες προτιμήσεις. Και εμείς είχαμε ταχθεί υπέρ του εμπορίου, των εμπορικών συναλλαγών ως αναπτυξιακή πορεία και οδό. Εάν δείτε το ποσό που προβλέπεται, εγώ βλέπω πώς ε, ισχύει και στην ΤΕΒΕ, βλέπουμε ότι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Ποιοι ευεργετούνται πραγματικά. Εγώ θεωρώ ότι με την οικονομική αυτή αρρωγή προς τις χώρες αυτές ε, δεν τις βγάζουμε από την φτώχεια, αλλά εάν προβάλλουμε τις εμπορικές συναλλαγές, τότε μπορούν να αποτάξουν το ζυγό της φτώχειας, διότι έτσι αυτές οι χώρες μπορούν να λάβουν αποφάσεις οι ίδιες και να προχωρήσουν κιόλας. Ίσως είναι δύσκολη η ερώτηση, αλλά όταν δίνετε χρήματα, δεν ξέρετε πού πάνε τα χρήματα. Θεωρητικά το ξέρετε. Έμπρακτα δεν μπορείτε να ιχνηλατήσετε την πορεία του χρήματος. Συμφωνώ βεβαίως ότι θα πρέπει να ε, γίνουν αυτές οι αναθεωρήσεις όπως και ο Κρίστοφερ. Πολλοί έχουμε αμφιβολίες για το ποιες χώρες πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και ποιες όχι. Θα ήθελα να υποβάλω ως τροπολογίες ως σημασίας. Εμείς γενικά ως ομάδα συμφωνούμε. Λάγκε. Σοσιαλιστές. Και δημοκράτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, συμφωνώ σε αυτό το θέμα με τον Ρόμπερτ Στέρντι. Το εμπόριο μπορεί να προωθήσει την ανάπτυξη, γι' αυτό θα πρέπει να διαμορφώσουμε έτσι και το αντίστοιχο σύστημα. Τι σημαίνει όμως αυτό. Τα κριτήρια για την ένταξη στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων θα πρέπει να γίνουν πιο αυστηρά. Διότι υπάρχουν χώρες που έχουν προχωρήσει αρκετά στην ανάπτυξη, οπότε ε, σιγά σιγά θα πρέπει να φεύγουν από το σύστημα. Ε, το πρώτο λοιπόν που θέλω να πω είναι τα κριτήρια, να κοιτάξουμε ποια είναι αυτά για να μπουν κάποιες χώρες στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Δεύτερον, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων συν. Σωστό είναι να έχουμε διευρυμένα κριτήρια για να κινούμε τις χώρες να έχουν βιώσιμη υφόρο οικονομία με κοινωνικές προδιαγραφές και πρότυπα. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ε, είναι και καλύτερη η έλεγχη. Ξέρουμε την υπόθεση με τη Σρι Λάνκα. Μετά από διαδικασίες ετών έχασε το καθεστώς της ένταξης στο GSP+. Θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν και να βελτιστοποιηθεί ο μηχανισμός παρακολούθησης και πώς μπορεί καλύτερα και περισσότερο να συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Και αυτό με φαίνει στο τρίτο μου για τις ασφαλιστικές δικλίδες. Με την Νότια Κορέα συζητήσαμε πάρα πολύ καιρό για τις ασφαλιστικές δικλίδες και διατάξεις και διευρύναμε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε αυτά και θα το ήθελα και στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. για να τονίσουμε ότι υπάρχει στενή συνεργασία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακριβώς για να βάζουμε και ασφαλιστικές δικλείδες σε αυτές τις συμφωνίες. Thank you, Ευχαριστώ Γιάννη Ξαντώ από τους Πρασίνους παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Φένε. Συμφωνώ και συμφωνώ και με τις επικρίσεις για τις δυσκολίες να ε, ορίσει κανείς τους καταλόγους και τα συγκεκριμένα κριτήρια. Εγώ θα είχα δύο συγκεκριμένα σημεία να θέσω που αφορούν κυρίως και απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, το Πακιστάν, ας πούμε, και οι Φιλιππίνες θα μπορούσαν να είναι επιλέξιμες χώρες στα πλαίσια του GSP+, αλλά τίθεται το εξής ερώτημα και σε σχέση με αυτά που είπε προηγουμένως ο Μπέρτ Λάγκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σταματήσει μόνο στην υπογραφή των διεθνών συμβάσεων και θα θεωρήσει ότι εντάξει το Πακιστάν για παράδειγμα ή άλλες χώρες σέβονται ε, μία σειρά δικαιωμάτων ή μήπως θα γίνει και καμιά έρευνα παρόλα αυτά για να κοιτάξουμε την πραγματικότητα. Λέω Πακιστάν, αλλά θα μπορούσα να σκεφτώ εδώ και τις δεσμεύσεις του Πακιστάν κατά της τρομοκρατίας. επίσημα είναι δεδομένες, αλλά στην πράξη ελέγχονται αυτές οι δεσμεύσεις κατά της τρομοκρατίας. Και επίσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει μια καταδικαστέα πρακτική, μεταξύ άλλων, που είναι η ιδέα να ε, αποσύρονται οι προτεμήσεις εάν μια χώρα επιβάλλει δασμούς στις εξαγωγές ορισμένων προϊόντων. Γνωρίζουμε ότι οι εξαγωγικοί δασμοί καμιά φορά μπορούν να βοηθήσουν ε, στην προστασία των φυσικών πόρων ή να προστατεύσουν ε, νεαρές βιομηχανίες και στην ανάπτυξη ε, αυτό είναι κατανοητό. Ο ΠΟΕ δεν καταδικάζει τέτοιου είδους εξαγωγικούς δασμούς. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι είναι αθέμητη πρακτική αυτή, unfair, ενώ μπορεί να εξυπηρετήσει στόχους αναπτυξιακούς. Μήπως είμαστε σε ένα σύστημα που προωθεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία περισσότερο και λιγότερο την ανάπτυξη των ελόγων κρατών. Ευχαριστώ. Ο Πολ Μέρφυ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τελευταία συζήτηση για το Ουσπεκιστάν μας δείχνει ακριβώς ότι δεν αρκεί να υπογράφει κανεί συμβάσει και συμφωνίε. Χρειάζεται ανεξάρτητη διερεύνηση των γεγονότων επιτόπου. Εδώ λοιπόν το κομβικό ζήτημα είναι τα κριτήρια. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αλλαγή κριτηρίων μπορεί να επηρεάσει εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους που θα χάσουν το καθεστώς GSP ή GSP Plus οι χώρες τους. Αρκεί να αναφέρει κανείς τον νησιμερινό και μόνο που θα βγει το GSP Plus με τα κριτήρια που προτείνονται τώρα. 350.000 ε, και εργάζονται στην αθοκομεία στο Ισημερινό, το 80% είναι γυναίκες. Και ε, δεν είναι μόνο η σημερινό και άλλες χώρες τη Λατινική Αμερικής θα πληγούν από αυτή την κατάσταση αν αλλάξουν τα κριτήρια. Ο Πρόεδρος. Προχωρούμε. Ωραία, προχωράμε. Στη θέση τη επιτροπή. Έχετε το λόγο. Θα ήθελα να υποβάλω κι εγώ μία ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έως και δύο Όταν μιλάμε για διαβάθμιση, η Επιτροπή άλλαξε τα κατόφλια έτσι ώστε όταν βλέπουμε τους αριθμούς θα είναι πιο δύσκολη η διαβάθμιση. Αλλά αυτό είναι απόρρια του γεγονότος ότι αφαιρέσαμε πολλές χώρες έτσι και για να, υπάρχει, να υπάρχουν ίδιες επιπτώσεις, το ίδιο αποτέλεσμα, θα πρέπει να αλλάξουμε τα κατόφλια για να υπάρχει η ίδια συμμετοχή στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων. Όμως υπάρχουν και τομείς, μάλλον ομαδοποιήσεις προϊόντων, που ε, είναι πιο περιορισμένες και θα πρέπει κανείς να είναι ε, πολύ πιο απόλυτος ε, ως προς τα κλωστοϊφαντουργικά, ας πούμε, για να είναι κανείς ε, ανταγωνιστικός. Δηλαδή θα πρέπει να μιλάμε για συγκεκριμένους τύπους υφασμάτων. Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο περιορισμός μάλλον αυτός ο υψηλότερος βαθμός ακρίβειας δεν κάνει και πιο δύσκολη τη διαβάθμιση, διότι αλλάζουμε κατηγορίες ε, προϊόντων. Και πώς, ε, πώς ισχύει αυτή η διάδραση με τη ε, διαβάθμιση. Δηλαδή πώς βγαίνουν ορισμένα προϊόντα και μετά υπάρχει νέα διαβάθμιση. Δηλαδή, αν υπάρχει υψηλότερη στοχοθέτηση, πώς έχει η διαβάθμιση και πώς βγαίνουν ορισμένα προϊόντα. Επίσης κάτι είπε ο Ρόμπερτ που με οδήγησε σε σκέψεις. Γιατί έχουμε μεγάλες και ωραίες ιδέες, αλλά ε, βλέπουμε ε, σε ορισμένες χώρες, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά Land Rover. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε σαφείς ως προς αυτή τη διαβάθμιση. Βεβαίως, οι εμπορικές συναλλαγές είναι καλύτερες από τη βοήθεια. Αλλά όταν μιλάμε για προτιμησιακό καθεστώς, ξέρουμε ποιες χώρες θα ευεργετηθούν από αυτές τις αφαιρέσεις. Ας πούμε ότι βγάζουμε τον Ισημερινό. Αυτό σημαίνει ότι ένας άλλος δικαιούχος των προτιμησιακών, των γενικευμένων προτιμήσεων θα προβεί σε εξαγωγές προς εμάς. Ή αν βγει ο Ισημερινός σημαίνει ότι αυτό το κενό θα το καλύψουν οι ΗΠΑ. Δηλαδή, αν πρόκειται για ανθοκομικά προϊόντα, αν αφαιρέσουμε δύο χώρες, ποιος θα μπει στη θέση τους, μήπως θα μπει ένας πλουσιότερος. Βεβαίως η Επιτροπή έχει κάνει εκατοντάδες χιλιάδες υπολογισμούς πριν φτάσει σε αυτό το σχήμα αλλά θα θέλαμε αυτή η ομαδοποίηση προτιμήσεων να μην χρησιμοποιηθεί από χώρες εκτός γενικευμένων προτιμήσεων, αλλά εντός γενικευμένων προτιμήσεων. Και τρίτη ερώτηση. GSP+. Ο κύριος Ζαντό μου υπενθύμησε ότι υπάρχουν δύο χώρες που θα προσθεθούν θα θεωρηθούν οι χώρες, οι Φιλιππίνες και το Πακιστάν, που θα πρέπει, για τις οποίες θα πρέπει να ισχύσουν οι κανόνες που προϋπάρχουν. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι χώρες έχουν κυρώσει τις συμβάσεις, αυτές τις 27 συμβάσεις ε, και το εποπτεύουμε αυτό. Ποιες είναι οι χώρες που θα μπορούσαν να κυρώσουν μία ή δύο συμβάσεις επιπλέον εάν τις πιέσουμε λιγάκι και να μπουν στον κατάλογο υποψηφίων χώρο. Γιατί στο GSP Plus έχουμε δύο νέες χώρες, αλλά θα ήθελα να γίνει τόσο δελεαστικό το GSP Plus, έτσι ώστε να έχουμε πέντε ή έξι υποψήφιες χώρες επιπροσθέτως και ποιες θα ήταν αυτές οι χώρες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι υπεψήφιες αυτό το GSP+. Πρόεδρος, θα ήθελα και εγώ να κάνω ορισμένα σχόλια πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Αυτό είναι κάτι το οποίο με απασχολεί και εμένα. Όταν μιλάμε για προτιμήσεις, μας ενδιαφέρουν, δηλαδή πρωτίστως ε, μας ενδιαφέρουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, δηλαδή επιχειρήσεις, καταναλωτές, αγρότες και οικονομικοί φορείς. Και τη στιγμή που υπάρχουν μονομερείς προτιμήσεις σημαίνει ότι έχουμε αδασμολόγητα προϊόντα από τρίτες χώρες. Δηλαδή μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά αυτά τα προϊόντα αδασμολόγητα και ανταγωνίζονται άλλες χώρες εκτός GPS. Και αυτό σημαίνει ότι ανταγωνίζονται τους δικούς μας εργαζόμενους, τις δικές μας επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Οι μονομερείς πρωτο, συμφωνίες τίθενται κατά του κανόνα MFN. Δηλαδή δεν υπάρχει ίση μεταχείριση τρίτων χωρών. Βεβαίως ο ΠΟΕ προβλέπει μία ε, ρήτρα ενίσχυσης, enabling clause, αλλά οι μονομερείς εμπορικές προτιμήσεις θα πρέπει να αποτελούν ένα έκτακτο πλαίσιο ως προς την κάλυψη. Κάλυψη γεωγραφική, κάλυψη προϊόντων και ούτω καθεξής. Εάν λοιπόν υπάρχουν τέτοιες γενικευμένες προτιμήσεις, τότε θα πρέπει να ζητήσουμε ένα αντάλλαγμα. Δηλαδή ε, να υπάρχει μια ρήτρα ερεσιμότητας. ως προς την κάλυψη αυτών των γενικευμένων προτιμήσεων. Δεν υπάρχει καμία τόσο αναπτυγμένη οικονομία με τόσο υψηλό προτιμησιακό καθεστώς όπως το GSP+. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε όταν ε, κοιτάμε την κάλυψη χωρών και μειώνονται οι χώρες, θα πρέπει το ευεργέτημα να στρέφεται προς τις πιο αναγκεμένες χώρες, δηλαδή τις ε, πλέον ενδεείς. και ως προς την αιρεσιμότητα θα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να κινηθούμε πέρα από την πρόταση της Επιτροπής. Δηλαδή να κινηθούμε πέραν. Οι μονομερείς ε, προτιμήσεις θα πρέπει να ισχύουν σε χώρες όπου ισχύει η θανατική ποινή, κάτι το οποίο δεν δεχόμαστε εμείς με βάση τις αξίες μας. Επίσης οι γενικευμένες προτιμήσεις θα πρέπει να ισχύουν ε, σε χώρες που δεν έχουν προσυπογράψει τη συμφωνία για τη μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Ε, επίσης όταν δεν έχουν συμφωνηθεί όταν δεν υπάρχουν συμφωνίες ως προς την κατάργηση της θανατικής ποινή, θα πρέπει να δεχτούμε αυτές τις χώρες. Έχετε πολλές ερωτήσεις, δηλαδή από τους κύριους Φιέλνερ, Στέρτη και από εμένα. Ο κύριος Φρανσίσκο Πέρες έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την αλληλεγγύη. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μας. Συνειδητοποιείτε πόσες δυσκολίες έχουμε για να καταλήξουμε σε μια πρόταση που να είναι ισορροπημένη και να επιτυχαίνει τους στόχους απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις, ε, αλλά γι' αυτό σας στέλνω και σας δείχνω αυτό το έγγραφο για να το δείτε, να δείτε και πώς φαίνεται. Τακτικά σας στέλνουμε επικαιροποιήσεις, ε, πακέτα πληροφοριών και ε, τις πιο συχνές ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους, με πολλές πληροφορίες. Είμαστε στη διάθεσή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα και ζητήματα, μην διστάσετε ποτέ να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα, ας πάμε στις ερωτήσεις σας και ξεκινώ με τι ερωτήσει του κύριου Μέρφυ. Φαίνεται να υποδεικνύουν ότι αν πρέπει να δούμε αν θέλουμε το εμπόριο και την αρρωγή ως δύο αντιφατικά ζητήματα. Πιστεύουμε ότι οι προτιμήσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τις ευκαιρίες για τις φτωχέ χώρες προς εξαγωγές και αν καταφέρουμε να επανεστιώσουμε την βοήθειά μας που να δίνει περισσότερη δύναμη, αφαιρώντας για παράδειγμα ε, περιορισμούς στις δυνατότητες, ε, δίνοντας διευκολύνσεις στο εμπόριο. Αν ε, δώσουμε αυτές τις ευκολίες στις φτωχότερες χώρες θα ήταν η ιδανική περίπτωση. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι ακριβώς αυτή τη στιγμή εμείς στην Επιτροπή επεξεργαζόμαστε ένα ανακοίνωθεν για το εμπόριο, για επενδύσεις και ανάπτυξη για να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε τις προτιμήσεις και την αρρωγή να συνδυαστούν έτσι ώστε να έχουμε ένα μέγιστο, βέλτιστο και αποδοτικό αποτέλεσμα. Τώρα, τέθηκαν αρκετές ερωτήσεις στο θέμα των κριτηρίων που προτείνουμε για να διαφοροποιήσουμε αυτές που δεν χρειάζονται ε, πραγματικά προτιμήσεις και αυτές που χρειάζονται. Θα ήθελα να προειδοποιήσω ε, λίγο ότι ο τρόπος που το έχουμε προσεγγίσει το θέμα είναι ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα κριτήρια είναι αντικειμενικά, αξιόπιστα και διεθνώς αποδεκτά. Γιατί, και θα ε, αναφερθώ και στον κύριο Μορέιρα εδώ, έχουμε νομικούς περιορισμούς στο πλαίσιο του νόμου του ΠΟΕ. Ε, έχουμε κάποιες δυνατότητες, αλλά ε, οι δείκτες μερικές φορές δεν ήταν αντικειμενικοί, δεν ήταν ολοκληρωμένοι και πλήρης δεν αφορούσαν τις διάφορες χώρες. Και ε, σε περαιτέρω συζήτηση αυτού του θέματος θα ήθελα να έχετε αυτό υπόψη σας. Τώρα το θέμα του GSP Plus και της παρακολούθησης. Στο σχεδιασμό αυτού του νέου κανονισμού έχουμε δει τα διδάγματα του παρελθόντος από τη διεύρυνση της Σρι για το ε, GSP+. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπήρχαν ελλείψεις στο σύστημα και είναι γι' αυτό που προσπαθήσαμε να τα δούμε σε όλα τα στάδια. Πρώτα, στο στάδιο όπου οι χώρες εισέρχονται στο σύστημα ένα μείζον πρόβλημα ήταν ότι δεν είχαμε ορίσει τι σημαίνει αποτελεσματική υλοποίηση και ήταν πολύ δύσκολο να κρίνουμε πώς να εφαρμόσουμε αυτά τα κριτήρια. Τώρα υπάρχει ο ορισμός μέσα στον κανονισμό Δεύτερο, υπήρχε ένα παραθυράκι όπου οι χώρε μπορούσαν απλά να ακυρώσουν την σύμβαση, αλλά με μια επιφύλαξη, για παράδειγμα, σχετικά με τη δυνατότητα του οργανισμού παρακολούθηση να κάνει τη δουλειά του. Αυτό είναι δυνατό στο νόμο αυτή τη στιγμή. Τώρα έχουμε αφαιρέσει αυτό το παραθυράκι. Έτσι, χώρε οι οποίε έχουν επιφυλάξει που μα εμποδίζουν στο έργο τη παρακολούθηση δεν θα γίνουν αποδεκτέ μέσα στο σύστημα. Αυτό για να σα δώσω μια μικρή γεύση. Βέβαια, αν αναρωτιέστε ε, αρκεί η απλή κύρωση, έχουμε προσθέσει μια τρίτη προϋπόθεση, δηλαδή ότι οποιαδήποτε χώρα η οποία ε, έχει σοβαρά ελλείμματα ε, στις αρχές της σύμβασης δεν θα μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα. Και αυτό βέβαια αντανακλά το θέμα ότι θέλουμε να είναι ένα σχέδιο που να βασίζεται σε κίνητρα. Καμία από αυτές τις χώρες δεν μπορεί να είναι όπως η Νορβηγία, αλλά με κίνητρα μπορούμε να δώσουμε τη δυνατότητα στις χώρες να φτάσουν επίπεδα. ένα επίπεδο. Επίσης έχουμε ενισχύσει την παρακολούθηση. Θα έρθουμε στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, θα ερχόμαστε όχι κάθε τρία χρόνια, αλλά κάθε δύο για να σας δείχνουμε τι κάνουν οι χώρες και το σημαντικό είναι ότι θα είμαστε στη θέση να χρησιμοποιούμε πηγές, όχι μόνο τις πηγές των φορέων και οργάνων παρακολούθησης που έχουμε αυτή τη στιγμή, αλλά και άλλες πηγές. Και αυτό είναι σημαντικό. Άλλες αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και αυτό επίσης φαίνεται ε, σε ένα μηχανισμό αποχώρησης που είναι πιο δυνατός, απόσυρσης που είναι πιο δυνατός από τον προηγούμενο που είχαμε τώρα. Το θέμα του αντικτύπου των τομέων. Έχουμε διαχωρίσει τις κατηγορίες των προϊόντων με διαφορετικό τρόπο, ε, με πιο λεπτομερή τρόπο αν θέλετε. Το θέμα είναι, αυτό θα οδηγήσει σε περαιτέρω διαβάθμιση. Δεν μπορώ να σας απαντήσω επί του θέματος. Δεν θα ήταν τίμιο εκ μέρους μου να το κάνω, διότι θα εξαρτηθεί από τις διάφορες ροές εισαγωγών από τις διάφορες χώρες. Αλλά ε, η επίπτωση που έχουμε δει από τους αριθμούς τώρα είναι ότι θα υπάρχει μία αποδιαβάθμιση για το Βιετνάμ για διάφορα προϊόντα βυρσοδεψίας είναι το μόνο στοιχείο που έχουμε. Ένα σημαντικό σημείο και ένα θέμα που αφορά το σημερινό. Ε, ο σημερινό εξακολουθεί να είναι μέρο του συστήματο. Είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να θέσω ευθαρσός. Όμως τώρα ο σημερινό είναι μια οικονομία ανώτερου μεσαίου εισοδήματος αν για τρει συνεχόμενες χρονιέ ο σημερινός διατηρηθεί σε αυτή την κατηγορία, τότε θα θεωρηθεί ότι δεν χρειάζεται, δεν χρήζει προτιμήσεων. Ε, υπογραμμίζω τις τρεις συνεχόμενες χρονιές, διότι καμία ε, χώρα δεν μπορεί μέσα σε ε, μια μέρα να εκδιωχθεί από το σύστημα. Θα περιμένουμε να δούμε αυτά τα τρία χρόνια, να δούμε αν υπάρξει αύξηση του εισοδήματος. Αυτό θα βοηθήσει. Η έξοδος των χωρών, δηλαδή από τον κατάλογο των διώχων, θα βοηθήσει αυτούς που έχουν πραγματική ανάγκη. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων δείχνει ότι ναι, θα υπάρχει σημαντικός επιπρόσθετος χώρος που θα δημιουργηθεί για άλλες ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες ε, για ε, να εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, είμαστε σε μια ενιαία αγορά ανταγωνισμός είναι ο κανόνας και δεν αποκλείεται άλλες χώρες να υποφεληθούν ε, οριακά. Δεν αποκλείω και ότι και οι θα έχουν κάποια πλεονεκτήματα οριακά. Αλλά αυτό είναι το σημαντικό. Για μας το σημαντικό είναι ε, ενώ προσφέρουμε περαιτέρω χώρο για αυτούς που χρειάζονται η αλλαγή στο σύστημα αξίζει τον κόπο. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν θα σας δώσω όλα τα τεχνικά στοιχεία της αξιολόγησης αντικτύπων, αλλά αν δείτε τα προϊόντα που εξάγονται από αυτές τις χώρες που δεν θα είναι πια δικαιούχοι και αυτές που παραμένουν, υπάρχει μεγάλη αντιστοιχία. Δηλαδή, ε, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να δημιουργηθεί επιπρόσθετος ε, ε, χώρος. Ένα τελευταίο σημείο ίσως τώρα που έχει να κάνει με την, την αιρεσιμότητα. Και ε, ε, έχω αυτά που είπε και ο κύριος Μορέρα. Είναι σημαντικό ότι ακολουθούμε τους κανόνες του ε, ΠΟΕ. Ε, και γνωρίζετε ότι ήδη δυστυχώς δεν είχαμε επιτυχία σε ένα πάνελ για ε, το σύστημα γυναικευμένων προτιμήσεων στο παρελθόν. Χάσαμε αρκετά στοιχεία στην υπόθεση. Ήταν ένα πάνελ ε, ε, που είχε φέρει η Ινδία σχετικά με το προκάτοχο του GSP+. Η ερασιμότητα είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα γιατί αυτό που μας επιτρέπει ο ΠΟΕ είναι να διαφοροποιήσουμε αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες εμπορίου, ανάπτυξης και επενδύσεων των δικαιούχων. Των δικαιούχων. Θα ήθελα να κλείσω εδώ και πάλι απευθύνω ε, έκκληση σε εσά, η πρόσκληση σε εσά να ε, επικοινωνείτε μαζί μας αν έχετε οποιασδήποτε ερωτήσεις θα είμαστε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Ο Κρίστοφερ Φιέλνερ για τα τελικά σχόλια. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ. Μου κάνει εντύπωση, μου κάνει εντύπωση, με ανησυχεί. Μου λέτε ότι βρίσκομαι στο σωστό δρόμο και δεν είμαι συνηθισμένος ε, σε κάτι τέτοιο. Τότε, αν όλοι συμφωνείτε, τότε κάτι πάει λάθος. Κάτι πάει καλά. Εν πάση περιπτώσει, ίσως να ισχύει αυτό και να μπορούμε να κινηθούμε εν αρμονία. Σε σχέση με κάτι που είπε ο πρόεδρος, ε, τώρα θα ήθελα να φτάσουμε σε ιδεολογικά ζητήματα. Γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Είπατε λοιπόν, η εμπορική μας πολιτική είναι, υπάρχει για την προάσπιση των δικών μας συμφερόντων και συμφωνώ. Συμφωνώ. Αυτό κάνουμε. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές για το ποιο είναι το κοινό συμφέρον, πώς μπορούμε να κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και ούτω καθεξής. Όταν μιλάμε όμως για GSP, δεν θα ήθελα να προσπιστούμε να προστατεύσουμε το δικό μας συμφέρον. Το GSP υπάρχει για να υποστηρίξουμε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω εμπορικών σχέσεων. Αυτό, αυτό, ε, αυτό, αυτή, είναι, ήταν η θεμέλια λήθος αυτού του σχήματος. Μετά, αν θέλουμε να συζητήσουμε τα δικά μας συμφέροντα, θα πρέπει να συντάξω άλλη έκθεση, δηλαδή για να πούμε τι κερδίζουν οι εισαγωγείς, τι κερδίζουν οι εξαγωγείς και ούτω καθεξής. Αυτό έχει σημασία, αυτό που έχει σημασία είναι κατά πόσο υπερασπιζόμαστε τις αναπτυσσόμενες χώρες. Έπειτα μιλήσατε πρόεδρε για μονομερείς προτιμήσεις. Ναι βεβαίως, το GSP ισχύει κάτι τέτοιο. Και ειλικρινά δεν θα ήθελα να υπάρχει αιρεσιμότητα και να ζητήσω ένα αντάλλαγμα, γιατί τότε δεν υπάρχει μονομέρεια. Μιλάμε για εμπορικές διαπραγματεύσεις και συναλλαγές και επειδή πρόκειται για φτωχές χώρες, θέλω να ζητήσω κάτι χωρίς ανταλλάγματα για το GSP. Για το GSP Plus το ζήτημα είναι διαφορετικό. Εκεί έχετε δίκιο, ας ζητήσουμε ανταλλάγματα, αλλά κάτι το πολύ συγκεκριμένο. Δηλαδή να συμπεριφερθούν σωστά αυτές οι χώρες. Να ισχύει το κράτος δικαίου, τα εργασιακά δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή να μην μιλήσουμε για ε, οικονομικά ευεργετήματα προς εμάς. Το μόνο αντάλλαγμα θα είναι πάλι κάτι το θετικό για τον κόσμο. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας ήπια ε, δύναμη μόχλευσης υπέρ του GSP+. Γι' αυτό και νομίζω ότι η Επιτροπή ανέφερε κάτι σημαντικό και ίσως θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτό είπε η Επίτροπη και αξιολόγησε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε χώρο για τις χώρες GSP, για τις χώρες που θέλουν αυτές τις ε, ε, γενικευμένες προτιμήσεις. Θέλω όμως να ξέρω κατά πόσο θέλουν να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλαίσιο, αλλιώς δεν θα έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, δηλαδή δεν βοηθήσουμε τις ε, λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα έχω ολοκληρώσει τη σύνταξη έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Και στις 8 Δεκεμβρίου να το ψηφίσουμε. Όποιος θέλει να πιούμε ένα καφέ, να το συζητήσουμε χαλαρά, είναι ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, 8 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε την έκθεση και θα ψηφίσουμε. 8. Εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα εξ ονόματο της Επιτροπής μας να καλωσορίσω τον κύριο Ντέιβιτ Πλάνκετ, ο οποίος βρίσκεται εκ δεξιών μου και ο οποίος είναι ο διορισμένος πρέσβης του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πρώτη φορά έρχεται στην Επιτροπή μας στο παρελθόν είχαμε εδώ μαζί μας τον προκάτοχό σας, τον κύριο Χόνμπι, καθώς και τον κύριο Φερχόιλ, που ήταν ο επικεφαλής εμπορικών σχέσεων στα πλαίσια της ΣΕΤΑ. Σας παρακαλώ μπορείτε να με ακούσετε. Λίγη ησυχία. Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο νωρίτερα φέτος ενέκρινε ένα ψήφισμα για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά. Εμείς παρακολουθούμε ματεύσει ΣΕΤΑ γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε πώς θα έχει έκβαση των διαπραγματεύσεων και για. αυτό αυτό ε, θα μεταβεί μία αντιπροσωπεία στον Καναδά μετά τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων και γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε πολύ πολύ καλό χρονισμό σχέσεων και επαφών στην Οτάβα και στο Τορόντο. Επειδή έχουμε 40 λεπτά στη διάθεσή μας για αυτό το θέμα, θα ήθελα να κάνετε μια αρχική δήλωση έτσι ώστε να αρχίσουμε τις συζητήσεις 15 λεπτά το πολύ και έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με καλέσατε ε, ενώπιον σας σήμερα Πρόσφατα έφτασα στις Βρυξέλλες να αναλάβω τα καθήκοντά μου και πρέπει να σας πω ότι είναι τιμή μου να διατελώ αυτή τη στιγμή ε, ε, στις Βρυξέλλες. Είναι πολύ ενδιαφέροντες καιροί και για τον Καναδά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις ε, μεταξύ μας σχέσεις και γενικότερα. Όπως γνωρίζετε προχωρούμε σε δύο σημαντικές διαπραγματεύσεις συνολική εμπορική και οικονομική σχέση και τη στρατηγική οικονομική ε, σχέση. Η ΣΕΤΑ ε, είναι ε, πραγματικά η κορονής ε, των συνομιλιών από τον Ιούνιο έχει θέσει πολύ μεγάλη προτεραιότητα σε αυτό η κυβέρνηση του Καναδά. Σε καιρούς οικονομικής αβεβαιότητας και ανασφάλειας η Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη με επενδύσεις και εμπόριο. Επίσης θα στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο ότι ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση απορρίπτουν τον οικονομικό προστατευτισμό και ανοίγουν τις αγορές. Εάν δύο χώρες βιομηχανικές, μάλλον δύο περιοχές, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς συμφωνήσουν, θα στείλουν ένα σαφέστερο μήνυμα στον υπόλοιπο κόσμο για το πόσο σημασία έχει η ε, περαιτέρω απελευθέρωση του εμπορίου. Επιπλέον, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, αν ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα βοηθήσει να προχωρήσουμε στις κοινέ μας δημοκρατικές αρχές. Θα ήθελα να πω ότι είμαι πάρα πολύ ε, ικανοποιημένο και χαρούμενος που αρχέ Νοεμβρίου ε, αποστολή τη Επιτροπής σα θα μεταβεί στον Καναδά, στην Οτάβα και στο Τορόντο για να καταλάβετε, να γνωρίσετε την οικονομία της χώρας μου. Επίσης, ε, είναι μεγάλη η προσήλωση και η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της κυβέρνησης, ε, της κεντρικής των επαρχιακών και τοπικών κυβερνήσεων, των επιχειρηματιών και γενικότερα των κλάδων της οικονομίας. Για τη συμφωνία ε, για την οικονομία και το εμπόριο, τη στρατηγική συμφωνία για την οικονομία και το εμπόριο. Γιατί η συνολική λοιπόν αυτή η συμφωνία ΣΥΤΑ από το 2010 ε, έχουμε 49 δισεκατομμύρια πλεόνασμα στις εξαγωγές μας και 55 δισεκατομμύρια είναι οι εισαγωγές ε, από την Ένωση Υπηρεσιών και Αγαθών. 146 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2010 και οι επενδύσεις ε, του Καναδά και 149 δις συνδυασμένες ε, επενδύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά. Σύνολο 294 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ισχυρός εταίρος ελκυστικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση με υγιή δημόσια οικονομικά. Βρισκόμαστε σε μια ισχυρή δημοσιονομική κατάσταση και επωφελούμαστε από ε, υγιή ε, δημοσιονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα. Οι τράπεζες είναι καλά οργανωμένες, με πολλά κεφάλαια, με καλή εποπτεία και μεγάλη διαφοροποίηση. Το Forbes ε, μας όρισε ως την υπαριθμό ένα χώρο στον κόσμο ε, για τις επιχειρήσεις με 11 παράγοντες, ε, καινοτομία, γραφειοκρατία, προστασία επενδυτών, αγορά και άλλους. Η, η Ένωση και ο Καναδάς το 2009 στην Πράγα ολοκλήρωσαν τι διαπραγματεύσει και αποφάσισαν να προχωρήσουν στη ΣΕΤΑ. Έχουν γίνει 8 γύροι και ακολουθεί ο ένατος προσεχώς με τρόπο επικοδομητικό συνεργαζόμαστε σε πνεύμα συνεννόησης και ακολουθούμε να εστιάζουμε και προσβλέπουμε σε μια επιτυχή έκφαση. Ήδη έχουμε ξεπεράσει και γεφυρώσει πολλές διαφορές. Και αυτό το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στους δύο επικεφαλείς εκατέρωθεν των διαπραγματεύσεων οι οποίοι σφυριλάτησαν ήδη αυτή την ατμόσφαιρα. Έχει προχωρήσει πολύ το κείμενο, έχει γίνει πρόοδος σε όλους τους τομείς και θα είναι ε, σημαντικός ο επόμενος και ένατος γύρος. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχιστεί στο ίδιο πνεύμα γιατί θέλουν να ολοκληρωθεί το έργο οι διαπραγματευτές το 2011. Οι επαρχίες και τα εδάφη του Καναδά επίσης ενδιαφέρονται πολύ να δοθεί ταχεία επιτυχής έκβαση. Παραμένουν προσιλωμένοι είναι και ορισμένοι τομείς που εμπίπτουν πλήρως ή στην ε, δικαιοδοσία τους. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Ξέρω ότι θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε τουλάχιστον μία επαρχιακή κυβέρνηση στον Καναδά για να καταλάβετε και μάθετε περισσότερο πόσο σημαντικό ρόλο παίζουν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Είναι πάγια και συνεχής η υποστήριξη των επιχειρηματιών για τη ΣΥΤΑ και για πιο μεγάλη σύσφυξη το δεσμό μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρούν διαπραγματεύσεις. Επίσης, ξέρω ότι θα δείτε και επιχειρηματίες ε, στον Καναδά. Σας καλώ να εκμεταλλευτείτε όσο μπορείτε, να γνωρίσετε τις επιχειρήσεις μας, να δείτε πόσο εκπληκτικές δυνατότητες και ευκαιρίες προσφέρουν. Η κοινωνία των πολιτών επίσης παίζει σημαντικό ρόλο, γίνονται διαβουλεύσεις για να ενημερώνονται οι Καναδοί για το πώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για τη ΣΥΤΑ. Επίσης, ε, τα μέσα ενημέρωσης δίνουν προσοχή και πολλοί ε, σύλλογοι οργανώσεις πολιτών ε, έχουν δραστηριοποιηθεί και αποφαίνονται. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας είμαι βέβαιος ότι θα έχετε επαφές με διάφορες οργανώσεις και οι διαπραγματεύσεις αυτές για τον Καναδά είναι πολυπλοκότερες και σημαντικότερες ε, από το 1992 που ολοκληρώσαμε τη ζώνη ελευθέρων συναλλαγών ναύτα με τη ΣΥΠΑ και το Μεξικό. Ε, ε, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε μια τέτοια συμφωνία με τις G8 θα προχωρήσουμε, θα αυξήσουμε την οικονομία, θα δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και θα απελευθερώσουμε περισσότερο το παγκόσμιο εμπόριο με τη συμφωνία μας αυτή. Τώρα για την άλλη συμφωνία, για τη στρατηγική εταιρική σχέση. Έχουμε διαπραγματευτική εντολή και οι δύο πλευρέ έχει αρχίσει η διαδικασία ε, διαπραγματεύσεων με πρώτο γύρο στην Οτάβα μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Ήταν σημαντική αυτή η πρώτη συνάντηση ε, για να θέσουν τα θεμέλια και τις παραμέτρους της εντολής τους και ε, πώς θα εργαστούν στο εξής. Στόχος για τη συμφωνία αυτή είναι σαφής να αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε αυτή τη φιλοδοξία γιατί γνωρίζουμε ότι οι σχέσεις μας πλέον είναι πάρα πολύ στενές, ε, πάρα πολύ αναβαθμισμένες και πάρα πολύ όριμες. Η πρώτη ε, συμφωνία διμερής έγινε το 1959. Έχει αλλάξει εκτοτέ και ο κόσμος, βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειαζόμαστε σύγχρονη συμφωνία για να έχουμε αποτελεσματικούς διμερείς ε, μηχανισμούς για να μας υποστηρίξουν. Πώς θα φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους. Εμείς θέλουμε μία πάγια και μόνιμη ε, σχέση και συμφωνία για το μέλλον να είναι ένα στρατηγικό κείμενο πλην σύντομο που θα συμφωνήσουν οι ηγέτες μας στην επόμενη σύνοδο κορυφής, θα διατρανώνουν τις κοινέ αξίες και το πώς θέλουμε να ε, τις προωθήσουμε παγκοσμίως. Συνεργασία λοιπόν ε, και σε θέματα διεθνούς ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Ένας μηχανισμός στη συμφωνία θα πρέπει να αντανακλά αυτά τα ισχυρά θεμέλια. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε και να βεβαιωθούμε ότι ε, θα διευκολύνει η συμφωνία αυτή τις ισχύουσες ή τι μελλοντικέ, να αποφύγουμε οποιαδήποτε επικάλυψη ή παράλληλε. Ε, συμφωνίες που ενδεχομένως να είναι τροχοπέδι εμπόδιο σε μελλοντικές μας σχέσεις. Είναι δύο προηγμένες κοινωνίες και οικονομίες ε, που ε, συνάπτουν ισχυρούς δεσμούς και σχέσεις και αναπόφευκτα υπάρχουν θέματα στα οποία διαφέρουν ε, οι απόψεις μας ή μπορούν να εμφανιστούν διχογνωμίες. Θα πρέπει να συνεργαστούμε με επικοδομητικό πνεύμα γνωρίζοντας τις διεθνείς επιπτώσεις που θα έχουν όλες μας οι αποφάσεις στα μεγάλα θέματα πολιτικής σχεδόν οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται με επιστημονικά στοιχεία και να ε, στηρίζονται σε γεγονότα. Αλλιώς μπορεί να οδηγηθούμε ε, σε πολιτική με λανθασμένες αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει προτάσεις. Ανησυχούμε όμως για μια ε, πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να τονίσω ότι εμείς δεν ε, είμαστε αντίθετοι με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Καθόλου θέλουμε να περιοριστούν οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων. Ε, το πετρέλαιο ε, που παράγει ο Καναδάς, ε, το αργό ε, πετρέλαιο έχει αμφισβητηθεί, αλλά αυτό δεν είναι βάση επιστημονικών στοιχείων. Από το 1990 μέχρι το 2009 έχουν μειωθεί κατά 29% οι εκπομπές του καναδικού πετρελαίου, το βαρέλι σε αέρια του θερμοκηπίου και καυσαέρια γενικότερα. Είναι πολλές οι ε, ευρωπαϊκές εταιρείες που εργάζονται στον Καναδά και η ασφαλτούχη ε, άμοι είναι μια ε, πηγή παραγωγής καλού καυσίμου. Εμείς δεν αμφισβητούμε, επαναλαμβάνω, τους στόχους οδηγίας, αλλά δεν θέλουμε να είναι εις βάρος της οικονομίας του Καναδά. Επίσης, τα προϊόντα φώκιας ε, μας λυπεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι πραγματικά πολύ ε, μεγάλη η προσοχή μας, η επαγρύπνηση, η προστασία των ζώων, παράγονται τα προϊόντα αυτά με πάρα πολύ σωστό τρόπο και ε, προστατεύεται και η υγεία των ανθρώπων και η υγεία των ζώων. Είναι διαφορετική η προσέγγιση μας, αλλά θα πρέπει να συνεννοηθούμε, να φτάσουμε σε μία ε, κατάληξη πάλι με βάση επιστημονικά στοιχεία να μην περιορίζεται το εμπόριο περισσότερο από ό,τι πρέπει και να αντανακλάται η σημερινή πραγματικότητα και η γνώση. Ξέρουμε ότι είναι περίπλοκες οι σχέσεις μας. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχουν και διχογνωμίες και διαφωνίες, αλλά δεν θα πρέπει να διασαλεύσει αυτό τις διμερείς μας καλές σχέσεις. Επίσης πρέπει να σας πω ότι είμαστε προσιλωμένοι στη συνεχή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να φέρουμε σε αίσιο πέρας τις συμφωνίες αυτές, τη ΣΥΤΑ και τη ε, Συμφωνία εταιρική Σχέσης. Ο Καναδάς θέλει να συνεχίσει τη στενή συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τις επιτροπές του και τους βουλευτές. Προσβλέπουμε στη μελλοντική σας ε, επίσκεψη και θα χαρώ να σας εναντήσω προσωπικά. Σας εύχομαι καλή και ενημερωτική αποστολή στον Καναδά. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω ενώπιό σας και θα απαντήσω με χαρά σε οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Σας περάσουμε στα μέλη αυτής της Επιτροπής, ξεκινώντας με τον ε, μόνιμο εισηγητή μας, γιατί έχουμε μόνιμους εισηγητές τώρα για ε, τους ε, πλήστους εταίρους μας και ο μόνιμος εισηγητής είναι ο Κίτερ Στάσουνη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον οριστέντα Πρέσβη. Καλώς ορίσατε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας εύχομαι καλή τύχη στις ε, προσπάθειές σας ε, και ε, σύντομα πιστεύω θα εξαφανιστεί ο όρος οριστής περέσβης και θα αναλάβετε πλήρως τα καθήκοντά σας και θα, με την πλήρη συμμετοχή σας στην Συμφωνία ΣΕΤΑ και στην στρατηγική Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως ανέφερε και ο Πρόεδρος, έχω οριστεί ως εισηγητής για την Συμφωνία ΣΕΤΑ και θα συνομιλούμε, θα συνεργαστούμε συχνά αναμένω και το αποτέλεσμα ε, πιστεύω ότι θα είναι κάτι το πολύ, πολύ θετικό για αμφότερους γιατί ουσιαστικά συμφωνώ πλήρως με τα εισαγωγικά σας λόγια. Έχουμε πολλά να πετύχουμε και για τις δύο πλευρές και ε, περνάμε από πιο εύκολους, θετικούς σε πιο δύσκολους τομείς. Ε, ίσως να υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις σε κάποια θέματα, αλλά ελπίζω ε, τα, τα ζητήματα να επιληθούν όσοι είχε προγραμματιστεί ε, στην αρχή ε, στις ε, αρχή όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την ΣΥΤΑ και τις ε, συμφωνίες, τις εμπορικές συμφωνίες. Έχετε αναφερθεί και είναι μια ερώτηση σε ένα από τα πιο ευαίσθητα θέματα, στα θέματα των πετρελαιοφόρων άμμων και των προϊόντων φώκες και θέλω να τονίσω ότι συμφωνώ πλήρως ε, ότι αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο, στην τελική θετική έκβαση της Συμφωνίας ΕΤΑ. Οι άλλοι τομείς που εμπεριέχονται και που ελπίζω να επιληθούν στον επόμενο γύρο ο οποίος ξεκινά την επόμενη εβδομάδα και ε, είπατε ήδη ότι η αντιπροσωπεία μας θα βρίσκεται στον Καναδά στο τέλος του μήνα και θα είναι σε θέση να συνεισφέρει με την διαβούλευση και την συζήτηση να συνεισφέρει στην τελική έκβαση για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Διότι ήδη έχω πάρει κάποιες αρνητικές απόψεις που πιστεύουν μερικοί ότι παρατείνεται η διαδικασία, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ ε, πραγματικά δεν το βλέπω και θα είμαι έτοιμος να προσθέσω και να συμβάλλω όσο μπορώ για να κλείσει αυτή η συμφωνία το συντομότερο δυνατόν. Γιατί όπως είπατε κι εσείς, θέλουμε να παρέχουμε στον υπόλοιπο κόσμο ένα παράδειγμα που να δείχνει ότι ο οικονομικός προστατευτισμός δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος λειτουργίας και ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια που ζούμε τώρα και τα τελευταία τρία χρόνια αυτές οι οικονομικές συμφωνίες βοηθούν στην τόνωση της μεγέθυνσης της οικονομίας, του τομέα της απασχόλησης και μας φέρνουν τον ένα πιο κοντά στον άλλο, μας κάνουν πιο παραγωγικούς και συνεισφέρουμε στο παγκόσμιο εμπόδιο και στην παγκόσμια ανάπτυξη αλλά και γενικά στην ανθρωπότητα και τη δημοκρατία γιατί ε, έχουμε τις ευθύνες μας και ο Καναδάς, είπα και άλλες ε, μεγάλες δυνατές αναπτυγμένες χώρες ε, έχουν να κάνουν τη δική τους συνεισφορά και έχουν τις δικές τους ευθύνες, το δικό τους μερίδιο ευθυνών για την σταθερότητα στον κόσμο και την αύξηση και ενίσχυση της δημοκρατίας. Ελπίζω κάποιοι συνάδελφοι να έχουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Εγώ είμαι ευτυχής με αυτά που άκουσα από εσά και προσβλέπω στο κλεισμό της συνεργασίας μαζί σας. Καλώς ορίσατε και πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ. Um, uh, ευχαριστώ τον μόνιμο εισηγητή, τώρα Σκιόδης. Ε, ε, οι μόνιμοι συγητές ε, έχουν προτεραιότητα. Η κυρία Κοχμαρίν από την ομάδα των φιλελευθέρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να συζητήσετε μαζί μας και ευχαριστώ για αυτή την πολύ σαφή ειλικρινή και διαφανή παρουσίαση των συνεχιζομένων διαπραγματεύσεων. Γνωρίζετε ότι το Ευρωκοινοβούλιο από την συνθήκη της Λισαβόνας ε, θα πρέπει να εγκρίνει αυτού του τύπου τις διεθνείς συμφωνίες. Και είναι σημαντικό το γεγονός ότι παραβρίσκεστε εδώ και μας πληροφορείτε για τις συνεχιζόμενες ε, διαπραγματεύσεις ε, εδώ στην Επιτροπή ΙΝΤΑ της Ευρωπαϊκής, του, του Ευρωκοινοβουλίου. Γιατί έτσι είναι η διαδικασία. Είναι σαφέ σε όλου μα εδώ ότι η συμφωνία είναι ζωτική σημασία, είναι σημαντική και για την ΕΕ και τον Καναδά. Ο Καναδά είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό εταίρο, εμπορικό εταίρο, ό,τι αφορά τη βιομηχανία, τι υπηρεσίε, τα γεωργικά προϊόντα, όλου του τομεί. Είναι ε, σημαντικό να έχουμε μια γερή ε, συμφωνία με το πέραστον των διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σα τη διαφάνεια που έχετε επιδείξει. Το θέμα τώρα των προϊόντων φώκια και τη απαγόρευση. είναι ένα θέμα πολύ ε, κοντά στην καρδιά των ε, πολιτών και των εκπροσώπων των πολιτών της Ευρώπης. Πρόσφατα είχα να κάνω ένα ξεκαθάρισμα στο σπίτι των παππούδων μου και είχα βρει μια αναφορά από την δεκαετία του 70 στα τότε μέλη του Ευρωκοινοβουλίου για την απαγόρευση των προϊόντων φώκες. Και τα περισσότερα από τα μέλη ε, που βρίσκονται εδώ ίσως να θυμούνται εκείνη τη φουσκωτή φώκια που είχαμε μπροστά στην αίθουσα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Ε, όπως βλέπετε είναι κάτι το οποίο έχει την προσοχή των πολιτών και των ε, αποφασίζοντων σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Και εγώ φοβάμαι ότι στις εμπορικές ε, σχέσεις, ένα από αυτά τα σημεία μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα εάν δεν βρούμε κάποιο συμβιβασμό ε, και ε, αν δεν έχουμε την συμφωνή γνώμη και το Ευρωκοινοβουλίου. Βλέπω να ανέβει ο Πρόεδρος. Κλείνω εδώ και σας ευχαριστώ και πάλι. Μάλιστα, γιατί αρχίζει να πιέζει ο χρόνος. Παρακαλώ δύο λεπτά έκαστος στο εξή. Ο Ρόμπερτ Στέρντι που είναι σκιώδης συζητητή της ομάδας συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Σας ευχαριστώ ε, εξοχότατε. Δύο ερωτήσεις έχω τις εξή τρεις, πολύ σύντομα. Βέβαια αυτό θα ήταν ίσως καλύτερα μια ερώτηση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θα ήθελα να μάθω πώς έχει κατάσταση με τη Συμφωνία Πλαίσιο που είναι ε, αντικείμενο παράλληλης διαπραγμάτευσης, η πολιτική πτυχή παράλληλα με τη ΣΥΤΑ. ΣΕΤΑ. Η, κυρία Κοχμερίν και εγώ μπορεί να διαφωνούμε λίγο για τις φώκες. Είχα περάσει μια εβδομάδα με μια οικογένεια Ινουίτ και είδα στο βορρά εκεί που ζουν πώς προστατεύουν το περιβάλλον. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να προστατεύει έτσι το περιβάλλον. Και η γεωργία ήταν ένα καθόδες θέμα. Χαίρομαι που προωθείτε. Βεβαίως μην το πείτε στην Επιτρογή Γεωργίας, αλλά πάμε για ελεύθερη ε, αγορά. Αλλιώς ε, στα γεωργικά προϊόντα μπορεί να, και να σας πυροβολήσουν στο Κοινοβούλιο, άμα τους το πείτε. Ε, Πώς ε, ε, προχωρούν εκεί τα θέματα. Είναι ε, τεράστια η πρόοδος που γίνεται στα γεωργικά προϊόντα. Θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο. Ο Ντέβιτ Μάρτιν, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Uh, uh, um, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Ε, ευτυχώς βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει η πολιτική με την αλλαγή φρουρά, την αλλαγή του πρέσβη δηλαδή, της θέσης αυτής. Μιλήσατε για ε, βλάβη, για ζημία στο περιβάλλον σε σχέση με την χρήση ορισμένων ε, ουσιών και πιστεύω ότι η, α, ως προς τη χρήση αυτής της ε, πισούχας άμμου θα μπορούσε να έχει ε, ολέθρια αποτελέσματα. Τώρα, σε σχέση με θέματα εισαγωγών και προϊόντα φώκιας, δεν θα πρέπει να γίνονται εισαγωγές. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να φτάσουμε σε μία συμφωνία ε, ελευθέρων συναλλαγών με τον Καναδά και όπως ξέρετε υπήρχε μία διαφορά σε επίπεδο ΠΟΕ για το θέμα των εισαγωγών προϊόντων φώκιας. Και θα ήθελα να πω για τους Ινουίτ ότι αποκλείονται από αυτή την, εξαιρούνται από αυτή την απαγόρευση ε, προϊόντων φώκιας. Σε σχέση με τα φαρμακευτικά σκευάσματα, από τις πληροφορίες που έχω, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο οι προδιαγραφές πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με τα φαρμακευτικά σκευάσματα θα αυξήσει το κόστος φαρμάκων στον Καναδά. Ε, αν ναι, γιατί ε, υπάρχει αυτή η πληροφορία που εντάσσεται μέσα στα πλαίσια της εντολής διαπραγμάτευση. Από την Γκουε. Σόλτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τον κύριο Πρέσβη και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία και τις συζητήσει για μια μελλοντική εμπορική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά με τον ίδιο τρόπο. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μερικές ερωτήσεις που αφορούν την οικονομική συνεργασία με την ευρύτερη έννοια που αφορά η εμπορική συμφωνία. Ε, από αυτή την έννοια θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο εξή. Την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον περιβαλλοντικό κανονισμό. Δηλαδή έχουμε ένα στάνταρ εργαλείο για προστασία του περιβάλλοντος ως ε, στοιχείο του κοινοτικού κεκτημένου. Εσείς έχετε πάρα πολύ ψηλέ προδιαγραφές και προστασία για θέματα δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών κτλ. Και οι δύο πλευρές λοιπόν ως αναπτυγμένες ε, οικονομίες έχουν ε, μέσα προστασίας ε, της ζωής των πολιτών. Εσείς πώς θα βεβαιωθείτε ότι αυτή η συμφωνία θα καλύψει και δεν θα διαταράξει αυτά τα υψηλά επιτεύγματα που έχουμε κατέρωθεν. Γιατί είναι και αυτό αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην εμπορική πτυχή. Και επανέρχομαι στις ε, πισούχες άμμος. Ε, εγκρίθηκε η οδηγία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ποιότητα των ε, καυσίμων. Στις 5 Οκτωβρίου ο Καναδάος, όμως δήλωσε ότι θα διαπαρτηρηθεί και θα την καταγγείλει αυτή την οδηγία στον ΠΟΕ. Θα προσφύγει σε περίπτωση που εγκριθεί. Εσείς τι λέτε, αυτό το θέμα των άμμων που των ασφαλτούχων θα διαταράξει ε, το θέμα και τις διαπραγματεύσεις ε, στη ΣΕΤΑ και σε ό,τι αφορά ε, την αντιπροσωπεία στο Καναδά γερουσιαστής Τζον Φρέιζερ είπε ότι θεωρεί ότι οι βουλευτές οι κοινοβουλευτικοί δεν συμμετέχουν αρκετά στη διαδικασία συνοδείας της διαπραγμάτευσης και πλαισίωσης. Δεν είναι γερουσιαστής βέβαια διαπραγματευτής αλλά θα δούμε και τι λέει η κοινωνία των πολιτών. Ε, από την Ευρώπη της ε, Ελευθερίας και Δημοκρατίας ο σκαλισηγητής. Ε, συγχαρητήρια εξοχότατη για το διορισμό σας. Μερικές παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε. Είπε ο πρέσβης επανειλημμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να του θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι χώρα. Αποτελείται από 27 ξεχωριστές χώρες μέλη Πολλοί εδώ γύρω στις Βρυξέλλες θα ήθελαν ε, κάτι διαφορετικό, θα επιθυμούσαν, αλλά απλούστατα δεν έχουν τη δημοκρατική εντολή και ε, με τη μορφή που σήμερα υπάρχει δεν πρόκειται να το πάρουν ποτέ. Και θα ήθελα να πω και κάτι στην κυρία ε, δόκτωρα Κοχμερίνα, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο κύριος Φέλνερ μίλησε για τις εμπορικές συμφωνίες ως τρόπο ε, ανάκλασης και Η ήπια δύναμη. Η ομάδα μου διαφωνεί. Το εμπόριο είναι εμπόριο, πρόκειται για αμοιβαία ευημερία, είναι συμφωνία για αμοιβαίο εμπορικό συμφέρον και όφελο και δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε ως μέσα άσκησης ή ε, προβολής ε, των διαφόρων πολιτικών σκοπιμοτήτων ορισμένων. Καταλάβατε κύριε πρέσβη τι εννοώ Μπορεί να μην το ξέρουν πολλοί, αλλά η Βρετανία είχε εμπορική συμφωνία με τον Καναδά. Στη διάσκεψη της Οτάβας ήδη από το 1932 και χάσαμε αυτή τη συμφωνία μας το 1975 όταν μπήκαμε τότε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. σε αντίθεση με, από αυτά που λένε πολλοί ε, συνάδελφοι, από πλευράς εμπορικής η Βρετανία ε, πλήττεται ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεν χρειάζεται να τονίσω. Ε, μας είπατε ότι ε, έχουν αρκετά κεφάλαια οι τράπεζες και αρκετή ρύθμιση στον Καναδά. Καλή ρύθμιση λοιπόν και καλή κεφαλαιοποίηση. Θα λέγατε τίποτα από τα δύο αυτά για τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου χώρας ο Πρόεδρος. Δεν έχουμε χρόνο και θέλω να σας πω ε, ενημερωτικά ότι είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον το εμπόριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει προσυπογράψει αυτές τις συμφωνίες και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας μπορεί όποια χώρα θέλει να, να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πολ Μέρφυ. Ευχαριστώ τον ε, πρέσβη ο οποίος παρευρέθηκε εδώ. Θα ήθελα να το προβάλλω ε, μία ερώτηση για την ε, πράξη του, την ενεργειακή, την πράξη του Οντάριο για την ενέργεια. Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες είναι οι επιπτώσεις της διαπραγματεύσης ΣΕΤΑ. Θα πρόκειται για μία πράξη η οποία δεν είναι καθόλου φιλική η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του Καναδά θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να προωθηθεί, διότι δεν μπορούσε να παρέμβει η ίδια κατά αυτής της πράξης, της πράξης του Οντάριο για την ενέργεια. Και σε σχέση με την απαγόρευση προϊόντων φώκιας θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει και για το πόσιμο νερό ως προς τις διαπραγματεύσεις ΣΕΤΑ. Έχει απαντήσει η Κομισιόν. Επίσης, οι ε, δημόσιες προμήθειες ε, αφορούν και μεταφορά υδρογονανθράκων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, η αξιολόγηση, η μελέτη αξιολόγησης για το περιβάλλον θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις ε, αρνητικές επιπτώσεις. Όμως η Κομισιόν προωθεί το ζήτημα. Ποια είναι η θέση της καναδικής κυβέρνησης. Η κυρία Γέγκελ, που είναι αντιπρόεδρος της μόνιμης αντιπροσωπείας με τον Καναδά. Έχετε το λόγο κυρία Γέγκελ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γέγλε για τη δυνατότητα που μου δίνετε κύριε Πρόεδρε ως Αντιπρόεδρος αλλά και ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας αγαπητέ Ρόμπερτ όπως το γνωρίζεις δεν χρειάζεται να πυροβολούμε ένα τον άλλον ε, μπορεί να μην έχουμε την ίδια άποψη για όλα τα θέματα αλλά αυτά τα χρόνια συνεργαζόμαστε πολύ στενά ευχαριστώ πολύ εξοχότατε πρώτα για την παρουσία σας εδώ από τόσο πρώιμο στάδιο και επίση μπορείτε να αναγνωρίσετε από τη συζήτηση ότι έχει σημασία το γεγονό ότι είστε εδώ και έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε και να ακολουθήσουμε αυτή την ατραπό μαζί. Είναι διμερεί οι εμπορικέ συμφωνίε αυτέ, γιατί δεν προχωρεί ο ΠΟΕ και η Ντόχα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπου για να προχωρούμε με χώρε, να δρούμε, να κάνουμε εμπόριο, να βοηθούμε του ανθρώπου από κοινού και τι κοινωνίε. Τα κρίσιμα σημεία ακούστηκαν και είμαι από μια χώρα που ε, έχει πολλές δυνατότητες και επαφές και πρέπει να σας πω το εξής. Πήγα ε, με την αντιπροσωπεία και είδα πώς ε, γίνεται η εξόριξη πετρελαίου και από περιβαλλοντικές οργανώσεις άκουσα θετικά ως προς τις εξελίξεις και για την προστασία του περιβάλλοντος και στον Καναδά ότι προχωρά η υπόθεση. Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας παρακολούθησα όλη αυτή τη συζήτηση για τις φώκες. Και ξέρετε πραγματικά περί τίνων αριθμών πρόκειται. Ξέρετε ε, τι προβλήματα έχουν οι θάλασσες γιατί έχουν επίξει στη φώκια. Θα πρέπει να βρεθεί ε, άλλη μορφή ε, θύρας κυνηγιού της φώκιας και θα πρέπει να ξέρουμε όταν συζητάμε τέτοια πράγματα ακριβώς την κατάσταση και να μην βασιζόμαστε μόνο σε κάποια email διαφόρων οργανώσεων. Ε, σε αυτή την εμπορική συμφωνία λοιπόν, αν θέλουμε να βάλουμε στο επίκεντρο τόσο πολύ την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων, θα πρέπει σε πολλές άλλες συμφωνίες εμπορικές ε, να βάλουμε περισσότερο στο επίκεντρο και πολύ περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το κάνουμε, άρα δεν το κάνουμε. Λοιπόν, παρακαλώ να γίνεται ισόρροπη και η συζήτηση και η περισυλλογή στη συνέχεια. Και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσετε να πάρω το λόγο. Η Κάθριν Μπέρντα, η οποία δεν ήταν στον κατάλογο μου, ε, είχα σηκώσει το χέρι λίγο χρόνο πριν. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον πρέσβη, να τον συγχαρώ για το διορισμό του. Είμαι Βρετανίδα και έχουμε μεγάλη παράδοση ε, συνενετικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο, ο κύριος Ντάρτμουθ μίλησε για το Ηνωμένο Βασίλειο όμως πρόκειται για Ηνωμένο Βασίλειο, τέσσερις χώρες δηλαδή που βρίσκονται μαζί. Δεν ξέρω γιατί ε, δεν συνεργάζονται καλύτερα και όταν ε, προσχωρήσαμε, μπορέσαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσαμε να συνεργαζόμαστε πολύ καλύτερα ε, σε θέματα εμπορίου. Νομίζω, ναι, αλλά Είχαμε όμως ε, συμφωνία με τον Καναδά από το 1975. Δεν καταλαβαίνω. Συνεργασίας, μια συμφωνία συνεργασίας. Please. Uh, we are negotiating a trade agreement with Canada. Είχαμε συμφωνία από το 1932, την οποία χάσαμε ως το 1975. Έγινε μια παρέμβαση και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μιλήσατε για την πετρελαιοφόρο άμμο. Και νομίζω ότι θα πρέπει οι συμφωνίες μας να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν Πόσο φτάσαμε, πώς φτάσαμε σε συμφωνία σε σχέση με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων. Υπάρχει και το θέμα των προϊόντων φώκιας όπως προαναφέρθηκε ως προς τις υπηρεσίες υδάτων Το θέμα αυτό δείχνει ότι αφενός υπάρχει θέμα συζήτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων περιβάλλοντος και ε, σε σχέση με το Colombian Trade Agreement δεν ξέρω πώς μπορεί να συμπεριφερθεί. Ναι, αλλά τα τρία λεφτά ε, σχετίζοντα και την παρέμβαση του συναδέλφου. Θα ήθελα να μου πείτε πώς έχει το καθεστώς για το πόσιμο είδωρ. Ο πρέσβης έχει και πάλι το λόγο, έχετε μία σωρία ερωτήσεων, έχετε όμως όσο χρόνο θέλετε στη διάθεσή σας, όχι βέβαια και πάρα πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δέκα λεπτά σας αρκούν, λέει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο σύντομα μπορώ. Βέβαια υπάρχουν κάποιες λίγο δύσκολες ερωτήσεις. Μία μπορεί, μπορώ να απαντήσω ε, γρήγορα είναι το θέμα της συμφωνίας πλαισίου. Δηλαδή, κατά το πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων, οι δύο αντιπροσωπείες αποφάσισαν να αλλάξουν την ονομασία των διαπραγματεύσεων από Συμφωνία πολιτική ε, σε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας. Ε, εταιρικής σχέσης και ε, έχει αντικατασταθεί ονομασία, αλλά συζητείται, αλλά έχει απλά μια νέα ονομασία. Θα υπάρχουν και άλλα θέματα ονομασιών που θα αφήσω κατά μέρος για την ώρα. Το ΑΣΟ ό,τι την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων, θα ομαδοποιήσω τι απαντήσει εδώ. Όπως είπα, μας ανησυχεί το γεγονό ότι η Επιτροπή προτείνει να δώσει πλεονέκτημα στο αργό πετρέλαιο με ίδιο ή ε, υψηλότερες εκπομπές ε, θερμοκηπιακών αερίων. η ψηλότερε εκπομπες θερμοκηπιακων αεριων η δεν μπορεί να χειριζόμαστε την πυρελφόρο άμμο ω ε, διαφορετική. Οι ανεξάρτητε μελέτε έχουν δείξει ότι οι εκπομπέ είναι παρόμοιε ή χαμηλότερε από άλλα ε, αργά πετρέλαια ε, όπω αυτά από τη Βενεζουέλα, την Αγγόλα και την Ιγυρία. Και η σύσταση τη πυροελευθόρου άμμου δεν είναι μοναδική, το ίδιο όπω και άλλα, άλλες, άλλοι τύποι αργού πετρελαίου. Όπως είπα, υποστηρίζουμε το στόχο της μείωσης των εκπομπών θερμοκηπών, αλλά αν είναι αυτός ο στόχος θα πρέπει να δούμε ε, μια πηγή πετρελαίου που δεν είναι μέσα στην ε, προμήθεια της Ευρώπης. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιδιώκει να μειώσει την ένταση της προμήθεια καυσίμων θα πρέπει να δούμε ε, είναι τα αργά πετρέλαια τα οποία καταναλώνονται στην Ευρώπη και που συμβάλλουν στην αύξηση των εκπομπών. Ε, είμαι διατεθειμένος διότι το έχω κάνει πολλές φορές να αποδεχτώ ότι μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες και στην προετοιμασία μου έχω κάποιες πληροφορίες τις οποίες θα υποβάλω στην Επιτροπή που παρέχουν κάποια από τα στοιχεία και τους αριθμούς που πιστεύουμε εμείς ότι θα ε, μπορούν να υποβληθούν σε επιστημονικό έλεγχο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φώκες και πάλι δεν αποτελεί έκπληξη όταν ε, ήμουν στο Λονδίνο για δύο-τρεις εβδομάδες τον χρόνο είχα ε, έξω από την πρεσβεία διάφορους ε, να διαμαρτύρονται. Κατανοώ πληρώσει το πακέτο αυτό γιατί έχω βιώσει αυτό το θέμα από κοντά. Πρέπει να επενθυμίσω την Επιτροπή ότι η το κυνήγι ε, φώκες είναι μια νόμιμη δραστηριότητα και εφόρος ε, δραστηριότητα που παρέχει ε, πηγή τροφής για πολλές οικογένειες. Πιστεύουμε ο Καναδάς αποφάσισε να ε, ε, αμφισβητήσει την απαγόρευση. Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχουν ερωτήσεις για τη χρήση των δικαιωμάτων μας να το επιδιώξουμε στον ΠΟΕ, διότι όπως θα γνωρίζετε σε όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις, είτε είναι διμερείς ή πολυμερείς, χώρες που αναγνώρισαν ότι ακόμη και οι φίλοι διαφωνούν και υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης διαφορών για να επιληθούν αυτά που είναι συνεπή ή δεν είναι συνεπή. Είναι πολύ περίεργο ότι θεωρείται ως προσβολή να ε, χρησιμοποιηθεί ο ΠΟΕ για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Θα συνεχίσουμε να ε, υπερασπιζόμαστε την βιομηχανία των, της παραγωγής προϊόντων φώκες. Ε, όπως και σε όλες τις διμερείς ε, σχέσεις υπάρχουν σημεία στα οποία διαφέρουμε αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε αυτές τις διαφωνίες να ε, παρεμποδίσουν μια ισχυρή οικονομική εταιρική σχέση Σχέση και αυτό αφορά και το πρόγραμμα Ontario Fit είναι σημαντικό το, το πρόγραμμα του Ontario Fit οι διαβουλεύσεις έγιναν με τηλεδιάσκεψη στις 7 Δεκεμβρίου του 2011. Πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα του Οντάριο είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ και θα υπερασπιστούμε αυτού του προγράμματος. Αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι διαφωνίες ε, όπου χρησιμοποιείται ο ε, θα μπορούσαν να εμποδίσουν την, το κλείσιμο μιας ισχυρής οικονομικής εταιρικής σχέσης ανάμεσά μας. Για να δούμε πού είμαστε. Ναι. Είναι και αυτό ένα δημοφιλές ε, θέμα, το θέμα του ύδατος, του νερού. Έχω κάνει τις διαπραγματεύσεις, εμπορικές διαπραγματεύσεις με πολλές χώρες για πολλά χρόνια και κάθε τόσο επανέρχεται και το θέμα του νερού και συνήθως ε, είναι ε, εκπλήσει αυτούς από εμά που εμπλεκόμαστε σε αυτό τον τομέα γιατί ε, δεν καταλαβαίνουμε πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα. Είναι η θέση του Καναδά ότι το είδωρ στη φυσική του κατάσταση δεν θεωρείται ε, αγαθό ή προϊόν, άρα παραμένει εκτός του πεδίου εφαρμογή τη Συμφωνία Συμπορική Συμφωνία με τον Καναδά. Ε, τίποτα ε, μέσα στη συμφωνία αυτή δεν αποτρέπει τι ε, κυβερνήσεις κυβερνήσει να θέτουν πρότυπα για το ασφαλέ πόσιμο νερό. Στι διαπραγματεύσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσουμε να διατηρούμε το δικαίωμα κυβερνήσεων να παρέχουν υπηρεσίε υδατοπρομήθεια στου Καναδού. Η διανοητική ε, ιδιοκτησία, στο πλαίσιο της ΣΕΤΑ επίσης και με συγχωρείτε δεν μπορούμε να μπούμε στα λεπτομέρειες των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι είναι καλύτερο να το αφήσουμε στους διαπραγματευτές. Ε, μπορώ να μιλήσω έως ενός σημείου, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερο να το δείτε με τους δικούς σας διαπραγματευτές. Ε, μία συμφωνία ΣΕΤΑ θα ενισχύσει τις ε, εμπορικές σχέσεις αλλά και την ε, διανοητική ιδιοκτησία. Πιστεύουμε ότι η θέση μας σε αυτές τις διαπραγματεύσεις στηρίζεται στους δικούς μας ε, νόμους και πολιτικές και καθώς εξτάζουμε αυτό που διακυβεύεται στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει να ικανοποιηθούμε ότι οποιασδήποτε προτάσεις υποβάλλονται και οποιασδήποτε συμφωνίε ε, κλείνουν θα πρέπει να αντανακλούν και τα συμφέροντα του Καναδά. Ε, το σχετικά με το θέμα των φαρμακευτικών προϊόντων, ε, το θέμα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή ποιο θα είναι το μέρο τη τελική συμφωνία. Βέβαια, θα υπάρξουν κάποια προβλήματα με κάποιες ιδέες που έχουν υποβληθεί, αλλά αυτό είναι σύνηθε σε οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Το ίδιο ισχύει και αντίθετα. Σε κάθε διαδικασία διαπραγματεύσεων θα συνεχίσουμε να συζητάμε σε ε, κάθε περίπτωση που το θέμα διανοητικής ιδιοκτησίας αποτελεί ε, κεντρικό μέρο. Ε, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κλείσετε την παρέμβασή σας ε, το θέμα των κρατικών προμηθειών. Οι προμήθειες είναι μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων βεβαίως και, και έχουν γίνει ανταλλαγές ε, στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και θα δούμε πού θα, θα καταλήξουν τελικά στα πλαίσια ενός φιλόδοξου πακέτου. Κάποιος αναφέρθηκε στο ρόλο του Κοινοβουλίου. Σημειώνω ότι ε, εγώ υποστήριζα τις ε, συμφωνίες ελευθερού εμπορίου. Ε, είχα επισκεφθεί το κοινοβούλιο αρκετές φορές. Ξέρω ότι ε, διαπραγματευτής μας είχε παρευρεθεί στο κοινοβούλιο αρκετές φορές. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι σημαντικό μέρος της διατήρησης ενός υγιούς διαλόγου και συζήτησης με όλους τους εμπλεκόμενους ε, στα γενετικώς τροποποιημένα προϊόντα. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα για μας, αλλά θα πρέπει να επανέλθουμε με Συγκεκριμένε πληροφορίε, διότι οι απόψει μα για τα γενετικώ τροποποιημένα προϊόντα είναι διαφορετικές ε, και μπορούμε να σας δώσουμε εμείς κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για το θέμα αυτό. Δεν ξέρω αν έχω αφήσει κάτι πίσω. Όχι. Ε, Προσβλέπω στην ε, συνεργασία μας με την Επιτροπή εντός των επόμενων μηνών και με όλο τον σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη όταν ο, ο Καναδάς είναι ένα κράτος όπου το χόκι πάγου είναι πολύ σημαντικό και όταν είπα ότι θα ερχόμουν εδώ που συμμετέχει και ο Πίτερ Στάσνη μου είχε ζητηθεί να πάρω αυτόγραφα. Θα το αφήσω αυτή τη στιγμή βέβαια για την ώρα. Σας ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ που παρευρεθήκατε εδώ. Καλή τύχη λοιπόν στην ανάλυση των καθηκόντων σας ως ε, περέσβης ε, του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ακόμα και το σημείο 9 σχετικά με την τελωνιακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό το θέμα είχε δοθεί στην Επιτροπή ΙΜΚΟ λανθασμένα κατά την άποψή μου, διότι έχει να κάνει με το εμπόριο και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναθεώρηση του υπάρχοντος κανονισμού είναι για την ενίσχυση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής Ιδιοκτησία. όμως αποφασίσαμε να μην αμφισβητήσουμε την αρμοδιότητα της ΙΜΚΟ, αλλά ζητήσαμε για ενισχυμένη συνεργασία στο θέμα αυτό, ζητήσαμε για το άρθρο 50 του εσωτερικού κανονισμού, το θέμα ε, παραμένει ακόμη να αποφασιστεί εντός της ε, ΙΜΚΟ για το κατά πόσο ε, μπορούμε να έχουμε αυτή την ενισχυμένη συμμετοχή. Ο εισηγητής μας είναι ο Χωσέφαντρες Εφάντρας Μπαρέα και της δίνω το λόγο για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με αυτό που μόλι είπατε. Α ελπίσουμε αυτή η ενισχυμένη συνεργασία να δώσει μεγαλύτερη ε, σημασία το θέμα. Η έκθεση αυτή, ξέρετε, έχει δύο πτυχές. Μια οικονομική, διεθνούς εμπορίου και την προστασία του καταναλωτού. Ας επικεντρωθούμε στο διεθνές εμπόριο. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις, είτε αυτές είναι πολυεθνικές είτε είναι μικρομεσαίες. Για την ε, προστασία των σημάτων, απολέμηση της πειρατείας και των απομιμήσεων. Ε, είναι συντριπτικές οι στατιστικές πάνω από 80 ε, ε, ε, χιλιάδες κατασχέσεις έχουν γίνει με πάρα πολύ ε, μεγάλη αξία, πάνω από ένα δις ευρώ, με κύρια προέλευση την Κίνα. Είναι πολύ σημαντικό και για το ενδοκινοτικό εμπόριο, αλλά και για τις συναλλαγές ε, τις οικονομικές και τις εμπορικές συμφωνίες, προστασία των επενδύσεων, της αηφορίας, της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, την καινοτομία και την έρευνα τη στιγμή που χρειαζόμαστε εγγυήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των καταναλωτών. Οι προτάσεις που μπορούν να γίνουν είναι, για παράδειγμα, το άρθρο 2.5 πλαστά εμπορεύματα και απομιμήσεις εγώ θέλω να διατηρηθούν τα σήματα, λογότυποι, οι μάρκες και για να ενισχύονται οι τελεινωνιακοί έλεγχοι. Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να προχωρούν σε ένδικα μέσα γιατί αυτό ε, ισχύει σήμερα και είναι μεγάλο οικονομικό βάρος για τις μικρές επιχειρήσεις. Και οι περίφημες transit απομιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά εξαιρούνται θα μπορούσε να ενταχθεί προς το παρόν εξαιρούνται από τον κανονισμό και αυτό δεν μας φαίνεται σωστό. Θεωρούμε ότι η έκθεση είναι περίπλοκη. Ελπίζω να βοηθήσουν όλοι οι σκιώδες και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Είναι σημαντική η προστασία των δικών μας επιχειρήσεων που εργάζονται ε, νομοταγός και θα πρέπει να καταδιώκεται και να διώκεται και να τιμωρείται η μαύρη αγορά που τόσο πολύ πλήττει το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά να ακούσω τους συναδέλφους και όπως είπε και ο Πρόεδρος ε, ελπίζω να μάθω ποια είναι η δική μας αρμοδιότητα ακριβώ για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω άλλου και άλλα μέλη της Επιτροπής θέλουν το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι. Και περνούμε αμέσως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητήσαμε από τη Γενική Διεύθυνση Τάξουτ να στείλει κάποιο εκπρόσωπο στη συνεδρίασή μας. Δεν ξέρω αν παρευρίσκεται κανείς. Μπορείτε να συστηθείτε σας παρακαλώ. Η κυρία Καρολίν Εντρή. Σωστά τα λέω. Καλώς ορίσατε. Έχετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι επικεφαλής τμήματάρχης της ε, Γενικής Διεύθυνσης Tax Wood σε σχέση με τις ελέγχους στα τελωνία ε, για την προστασία των καταναλωτών σε σχέση με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι η Επιτροπή θα υποβάλει μία πρόταση. Ήδη υπάρχει ε, νομοθεσία σε σχέση με την ενίσχυση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στα σύνορα και θέλουμε να αντικαταστήσουμε την προϋπάρχουσα νομοθεσία έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε τα τελωνία να μπορούν να εφαρμόζουν την τήρηση των ε, πνευματικών δικαιωμάτων ε, εκτός συνόρων και επίσης να ξέρουμε ποιο είναι το, το διακύβημα όταν προωθείται κάτι τέτοιο. Όπως είπε λοιπόν και η συγγήτρια, θα πρέπει να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού έτσι ώστε τα, τα τελωνία να μπορούν να προβαίνουν στην κατάσχεση αγαθών όταν ε, παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας γιατί δεν είχαμε μπορέσει να καλύψουμε το παράλληλο εμπόριο μέχρι σήμερα, έξω από τα σύνορα. Επίσης υπάρχει ειδική νομοθεσία σε σχέση με την παραβίαση ε, των πνευματικών ε, δικαιωμάτων όταν πρόκειται για μικρές παρτίδες και αγαθά. Όταν πρόκειται λοιπόν για μικρές ε, ποσότητες, επειδή κρατούνται αυτά τα, τα προϊόντα, οι μικρές παρτίδες στα σύνορα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα την προστασία του καταναλωτή και μας απασχολεί και η τύχη αυτών των προϊόντων. Γι' αυτό μιλάμε για καταστροφή αυτών των προϊόντων, έγκαιρη καταστροφή αυτών των προϊόντων και πολλές φορές ε, ως προς τα γενώσιμα φάρμακα υπάρχουν διαφορές με την Ινδία ή τη Βραζιλία και θα θέλαμε να αποσαφηνίσουμε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τι θα πρέπει να κάνουν τα τελωνία όταν ε, βρίσκουν γενώσιμα φάρμακα σε διαμετακόμιση, σε τράνζιτ. Και Πώς τονίζουμε στο Μνημόνιο Συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ινδίας, τη στιγμή που υπάρχει διαμετακόμιση σκευασμάτων και τα γενώσιμα αυτά σκευάσματα προστατεύονται από τη δική μας νομοθεσία, δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι παραβιάζουν ε, πνευματική, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν υπάρχει υποψία ότι θα μπουν στην ευρωπαϊκή αγορά, τότε μπορούν να κατάσχουν αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωσέφα, τίποτα άλλο. Όχι, όχι, δεν έχω να κάνω καμία, καμία παρατήρηση. Στις 8 Δεκεμβρίου θα εξετάσουμε την έκθεση και θα υπάρξει ενισχυμένη συνεργασία με την ΙΜΚΟ επί του θέματος. Λοιπόν, λίγουν οι εργασίες μας ως προς την δημόσια συνεδρίαση του πρωινού. Τώρα έχουμε συνεδρίαση και κλεισμένο των θυρών των συντονιστών και θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από όλους όσους δεν μπορούν να παραμείνουν να αποχωρήσουν σύντομα και ήσυχα. Είπα σύντομα.